Συνάδελφοι, θα ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Να σας ρωτήσω αν μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Και επίσης έγκριση των πρακτικών. Είσαστε όλοι ικανοποιημένοι και με τα πρακτικά. Ωραία, συμφωνία περί υπηρεσιών του προχωρήσουμε στην συμφωνία περί υπηρεσιών του κυρίου Κοχ. Θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα ε, σπουδαστών μετάφρασης από το Λουξεμβούργο. Δεν ξέρω αν τους έστειλαν στην δική μας επιτροπή, επειδή θα είμαι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα απαντήσουν ε, στη σταδιοδρομία τους, ε, αλλά θα θέλαμε να τους καλωσορίσουμε. Έχουμε τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, σχετικά με ορισμένε πτυχέ των αεροπορικών υπηρεσιών του κυρίου Κοχ. Δίτερ, θα πρέπει να βγω για 5-10 λεπτά κατά τη διάρκεια ε, τη έκθεσή σου. Κανονικά θα ήσουν εσύ αντιπρόεδρο και θα έπρεπε να αναλάβει, αλλά επειδή είναι δική σου έκθεση, μήπω θα μπορούσα να παρακαλέσω Ποιος είναι επόμενος στη σειρά. Ε, ποιος μπορεί να προεδρεύσει πέντε λεπτά. Η κυρία Τιβέρακ. Μπορείτε παρακαλώ για πέντε λεπτά να αναλάβετε την Προεδρία. Ο κύριος Διγκράντες. Άμπλε παπλών θα κάνουμε. Ποιος θέλει να προεδρεύσει. Κριστίν, έλα. Για πέντε λεπτά μόνο. πρέπει να συναντηθώ με τον Ούγγρο πρέσβη. Η κυρία Τιβέρα, παρακαλώ. Donc je donne la parole à Monsieur Cork. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κόχ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με πολύ μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω σε εσά ιδιαίτερα την έκθεσή μου αλλά και στους συναδέλφους. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μία έκθεση που μου έπεσε ο κλήρος στα πλαίσια της ε, εναλλαγής ε, των εκθέσεων ε, είναι 47 ε, συμφωνίες μεταξύ των κρατών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της ε, Δυτικοαφρικανικής Νομισματικής και Οικονομικής Έκθεσης. Ε, ένωση, συγγνώμη. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Καστέξ και όλους που συνεισφέραν στην έκθεση αυτή. Ε, πρώτος στόχος της συμφωνίας αυτής ή των συμφωνιών είναι πρώτον η άρση των εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά και κατά δεύτερο λόγο η άρση και η κατάργηση των διατάξεων που δεν ανταποκρίνονται ε, στο επίκαιρο πλαίσιο ε, νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω ε, δρούν με διακρίσεις. Υπήρξε μια προσφυγή ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και αυτό οδήγησε και στις συμφωνίες γιατί υπήρξαν ε, μεμονωμένες παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Ένας επιχειρηματίας ή μια εταιρεία από μια χώρα της Ένωσης που ίδρυαν θηγατρική σε άλλη χώρα της Ένωσης δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτές τις συμφωνίες το Συμβούλιο προδικαστικά ήδη από το 2003 είχε δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, επανεξετάσει αυτά τις κρίσιμες διατάξεις ε, τις ε, προβληματικές να τις αλλάξει με την αρχή της χώρας προέλευσης. Πέρσι το Νοέμβριο 2009 υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία και εφαρμόζεται προσωρινά έκτοτε. Ε, σημαντικά αποτελέσματα ε, των διαπραγματεύσεων εκτός από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας ρυθμίστηκαν και μπήκαν και άλλα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου μεταξύ αυτών δυνατότητα φορολόγησης ενεργειακών προϊόντων ε, στις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις και καταργήθηκαν και οι προσαρμόστηκαν μάλλον άλλες ε, διατάξεις που στρέβλωναν τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα αναμένουμε να αρθούν και τα λοιπά εμπόδια για τη διάνοιξη της αγοράς. Στην εντολή Επίσης διαπιστώθηκε ότι ε, το κείμενο της συμφωνίας δεν αντιτίθεται με ε, την προσπάθειά μας για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Τροπολογίες μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Και την 1η Δεκεμβρίου, αν όλα πάνε καλά, θα ψηφιστεί η έκθεση στην Επιτροπή μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε με το Συμβούλιο ούτε με την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ανάβει αυτόματα για τον πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόχ για την παρουσίαση της έκθεσης. Να δώσω το λόγο στον κύριο Καντρονή. ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος για το θέμα αυτό. Μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση αυτή χωρίς καμία επιφύλαξη. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή ε, για το έργο του στο επόμενο θέμα θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις ε, για τις διεθνείς συμφωνίες εναέριων μεταφορών ε, που αυτά που θα πω ισχύουν και για το εδώ την έκθεση αλλά θέλω να τα αναφέρω στο επόμενο θέμα και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σχεδόν παρετείνει η συζήτηση διότι μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με τον ε, κύριο Ελχαντράουι. Ε, στις ε, συμφωνίες αυτές έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ναι ή όχι. Ο κύριος Κόχο εξήγησε πολύ καλά γιατί είναι χρήσιμο να στηρίξουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Για το επόμενο σημείο έχω κάποια πράγματα να πω, αλλά εδώ μπορούμε μόνο να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Πράτπορν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Η παρατήρηση του κυρίου Αρκαντράου για το επόμενο θέμα με βρίσκουν σύμφωνο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω ορισμένα σχόλια σε ό,τι αφορά τις γενικέ αρχέ που διέπουν αυτές τι συμφωνίε, αλλά πραγματικά συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη αυτή έκθεση από τον κύριο Κόπ. Pour la Επιτροπής, ο κ. Μπουργκελ Βερνέ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια για να πω ότι η Επιτροπή χαίρεται ιδιαίτερα με την έκθεση του κ. και με την προοπτική του να περατωθεί αυτή η συμφωνία. Όπως υπογράμμισε ο εισηγητής, είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία προσαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο με ορισμένε συμφωνίε, 47 συμφωνίε. Είναι επίση σημαντικό γιατί είναι η πρώτη συμφωνία αυτού του είδου που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα συγκρότημα χωρών, με μια ομάδα χωρών. Αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το υπογραμμίσουμε. Ευχαριστώ. Μήπως κάποιος θα επιθυμούσε να ξαναπάρει το λόγο. Ο κύριο Χοκ. Ε, ναι, με χαρά να ακολουθήσω αυτή την υπόδειξη, την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τη απουσία του Προέδρου όλοι είστε πάρα πολύ σύντομοι. Η ημερομηνια προθεσμιε προθεσμίες κατάθεση τροπολογιών 5η Νοεμβρίου για την ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών 1η Δεκεμβρίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια Ιανουάριο του 2011. Δυσκολεύομαι να συνεχίσω να προεδρεύω γιατί έχουμε τώρα την παρουσίαση της έκθεσης του κυρίου Σίμψον. Θα πρότεινα λοιπόν να διακόψουμε για λίγο μέχρι να έρθει ο πρόεδρος. Okay, ladies and gentlemen, sorry. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστώ πολύ, Κριστίν, που με αναπλήρωσες. Μόνο ότι στο είπα την τελευταία στιγμή. Τώρα, το επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης είναι η δική μου έκθεση. Μετά ανταλλαγή απόψε με η Βελική Προεδρία. Η κυρία Γέιγκερ έχει το λόγο από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Επιτροπής ε, θα ήθελα να πω ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου ενέκρινε μια νέα συμφωνία πλαίσιο που αφορά τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Ε, η συνθήκη τη Λισαβόνα ενδυναμώνει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι κάτι που αντικατοπτρίζεται στη νέα συμφωνία πλαίσιο. Εκτό από αυτό, η συμφωνία πλαίσιο είναι βασικό εργαλείο στην εφαρμογή τη νέα σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή. Η Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία απόφαση των εσωτερικών κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν του τρόπου ε, εφαρμογή τη συμφωνία πλαισίου. Συνεπώ, σήμερα δεν μπορώ να σας δώσω μια πλήρη απάντηση σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί απτά η Συμφωνία Πλαίσιο. Βεβαίως η Επιτροπή θα σεβαστεί όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, εννοείται, και θα εφαρμόσει τη Συμφωνία Πλαίσιο σύμφωνα με την ε, ιδιαίτερη σχέση που έχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοινοβούλιο η, αναφέρθηκε την Ολομέρα στις 16 Οκτωβρίου αυτό υπόθηκε ότι η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από κάποια μονομερή ερμηνεία της Συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση θα υπάρξουν καινοτομίε σε ό,τι αφορά το διαθροτικό διάλογο, τις συναντήσεις ειδικών, τους φορείς καθώς και τις διαπραγματεύσεις και τις διεθνείς συμφωνίες. Σε ό,τι αφορά το διαθροτικό διάλογο, ο Βητικάς θα υποβάλει ένα πρόγραμμα το 2011 στις 9 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα καταρχά να πω ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι οι συντονιστέ αποφάσισαν να συντάξουν μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία σχετικά με αυτό το θέμα. Θυμάμαι ότι στο παρελθόν το Κοινοβούλιο γνωμοδοτούσε μόνο για ορισμένε συμφωνίε. ενώ συχνά η γνώμη μας ήταν θετική, αυτό γινόταν με περιορισμένη συζήτηση. Βεβαίω, αυτές οι συμφωνίε απαιτούν την κοινοβουλευτική συνένεση. Θα πρέπει να τα δούμε, ε, ε, να εξετάσουμε κάπω πιο ενδελεχώ. Βεβαίω παραμένει η δυσκολία ότι η επιλογή είναι μεταξύ του ναι και του όχι, ακόμα και στι περιπτώσει τι πιο αντιφατικέ. συνεπώ η συζήτηση παραμένει περιορισμένη. Το που θα ήθελα να κάνω, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκθεση για να, να αναφερθώ σε δύο βασικά θέματα. Πρώτον, το περιεχόμενο των συμφωνιών και δεύτερον, το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και των, ε, της έγκρισής Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και την ουσία, πιστεύω ότι υπάρχει ευρία συνένεση ότι μία συμφωνία με τρίτε χώρες είναι κάτι θετικό. Βεβαίως οι οριζόντιες συμφωνίες που εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου του Νοεμβρίου του 2002 είναι αναγκαίες για να εξασφαλίσουν νομική βεβαιότητα. Επίσης εγγυώνται, εξασφαλίζουν τα ίδια δικαιώματα σε όλες τις αεροπορικές γραμμές της Ένωσης, ενώ από την άλλη πλευρά καλύπτουν τις συμφωνίες των χωρών μελών. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι γενικές συμφωνίες ε, με γειτονικέ χώρες <clears throat> μπορούν να οδηγήσουν σε ωφέλη και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά και την ποικιλία και το κόστος, παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες στις αεροπορικές εταιρείες. Εκτός από αυτό, η ρυθμιστική σύγκληση θα μπορούσε να συμβάλλει στην προώθηση του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι επιδοτήσει και το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστο. Θα πρέπει όμω να είμαστε προσεκτικοί, να μην πέσουμε στην παγίδα του να θεωρήσουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία είναι καλή συμφωνία. Αντίθετα, θα πρέπει να εξεταστεί ένα θέμα από την Επιτροπή ως διαπραγματευτή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως φορείς που θα πρέπει να εγκρίνουν το αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. Σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη συμφωνία είναι εξισορροπημένη και φιλόδοξη ή ενδεχομένω θα τα σκόπιμο να καθυστερήσουμε τη συμφωνία εν αναμονή ενός καλύτερου αποτελέσματος. Δεν θα ήθελα τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες αυτή τη χρονική στιγμή. Εάν εξετάσετε τις λεπτομέρειες της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, εδώ ο εισηγητής, ο κύριος Ζεζάντο, θα αναφερθεί σε αυτό το θέμα όταν μας υποβληθεί το αίτημα από το Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε στο ψήφισμα τη Ολομέρειας τον Ιούνιο, υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια σχετικά με την έλλειψη ισορροπία ό,τι αφορά τι ευκαιρίες επενδύσεων. Και από την άλλη πλευρά ε, ε, ε, θα πρέπει να σε ό,τι αφορά θέματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά να στοχεύουμε προς ψηλά και προς ε, χαμηλά. Θα πρέπει βεβαίως να αποφύγουμε την επικάλυψη των δοκιμών και των αξιολογήσεων εκτός βεβαίως αν υπάρχει μια σημαντική ρυθμιστική διαφορά και αυτό θα επιτρέψει τις, ε, τους κατασκευαστές να βασιστούν στο σύστημα πιστοποίηση. Ε, γιατί κάτι τέτοιο μας βοηθάει να επιτύχουμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Παρόλα αυτά η έκθεση σχετικά με τη συμφωνία με τον Καναδά που θα υιοθετηθεί αύριο αναφέρεται σε μερικές από αυτέ τι συμφωνίε, οι οποίε είναι πιο φιλόδοξε από άλλε. Είναι σημαντικό αυτέ οι συμφωνίε υψηλή ποιότητα να αποτελέσουν ένα υπόδειγμα για τι μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία ε, και την επιλογή ναι ή όχι, μόλις ε, περατωθεί η διαπραγμάτευση, ε, δίχως άλλο δεν έχουμε να κάνουμε με μια ιδανική κατάσταση. Όπως δείχνει η περίπτωση του SWIFT, Πολλέ φορέ με ένα όχι προσελκύει κανεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από το τύπο. Αλλά δεν φαίνεται να είναι μια στρατηγική που θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά. Κατά συνέπεια θα πρέπει να βρούμε τρόπου για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι η Επιτροπή θα γνωρίζει πώ θα αξιολογούμε μια συμφωνία πολύ πλήρη από τη λήξη τη σύναψη της συμφωνίας. Και ποιε είναι οι γραμμέ που θα μα καθοδηγήσουν. Βεβαίως αυτή δεν είναι μια καινούργια ιδέα. Ήδη μας έχει ενημερώσει η Επιτροπή κατά την προετοιμασία της ε, αντιπροσωπείας που πήγε στη Ουάσιγκτον τον Μάρτιο. Τίχως άλλο, αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να προβληματιστούμε. Η συμφωνία πλαίσιο με την Επιτροπή που συνήθι το 2005 δέσμευσε την Επιτροπή την παροχή έγκαιρων πληροφοριών στο Κοινοβούλιο και κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης των συμφωνιών και κατά τη διάρκεια της σύναψης ε, διεθνών, διεξαγωγής και σύναψης διεθνών συμφωνιών. Αυτό καλύπτει τις οδηγίες, το σχέδιο οδηγιών, τις ε, υιοθετημένες ε, οδηγίες, τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και την σύναψη αυτό και τη λήξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο κανόνας 90 παράγραφος 5 επιτρέπει στο Κοινοβούλιο με βάση μια έκθεση από την υπεύθυνη Επιτροπή να υιοθετήσει συστάσεις και να ζητήσει να ληφθούν υπόψη πριν τη σύναψη οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας. Το θέμα είναι το πόσο, τι, τι χρήση θέλουμε να κάνουμε αυτό. Τα σημεία που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι ότι υπάρχουν δυνατότητες που υπήρχαν πριν από την αναθεώρηση της ε, συμφωνίας και αυτές εγκρίσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό ενδυναμώνει τη δυνατότητα να εντατυχάνουμε όλοι οι ίσεις ε, αντιμετώπισης αλλά και της υιοθέτηση συστάσεων. Πριν να δώσω το λόγο στο σκιώδη συγητή, θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι περιμένω με ανυπομονησία να συνεργαστώ το μαζί τους για να καταλήξω σε μία συμφωνία. Η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι ένα σημείο εκκίνησης και με μεγάλη χαρά θα οργάνωνα άτυπες συνεδριάσεις όποτε παραστεί ανάγκη ή όποτε κάποιος το θελήσει. Με αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις θα έλεγα να περάσουμε στη συζήτηση έτσι ώστε να ενημερωθώ για την άποψή σας και αν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με βάση τα όσα σας είπα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τους συντονιστές. Όσον αφορά τη διαδικασία, είναι σαφές ότι πρώτον δεν θα πρέπει να ε, υπερτιμήσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Διότι η απόφαση αυτή είναι του τύπου ναι ή όχι. Και ξέρουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χάνονται πολλές αποχρώσεις. Και πολλοί συχνά το ναι υπερισχύει διότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ε, το κατά πόσο είναι απαραίτητο ένα όχι. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Ε, συμφωνούμε με αυτά που ε, συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο όσον αφορά Όσον αφορά το ύφο, ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι επειδή είναι σημαντικό το θέμα, θα πρέπει να πληρώσουμε και το αντίστοιχο τίμημα. Πιο σημαντικό για μένα είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Ε, το θέμα της ε, διαδικασίας συμφωνίας με την Κομισιόν και από τις δύο πλευρές θα πρέπει να υπάρχει βούληση και θα υπάρχει η υποχρέωση ενημέρωσης διότι συχνά είναι δύσκολο για μας, για το Κοινοβούλιο να καταλάβουμε τη διαδικασία ε, μιας συμφωνίας όταν δεν λαμβάνουμε εγκαίρως ε, τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης ε, δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε δομές όπου το Κοινοβούλιο ε, να συμμετέχει μέχρι τελευταία στιγμή. Ε, θα μπορούσε να το απαιτήσει κανείς, αλλά δεν ε, ξέρω πόσο χρήσιμο θα ήταν κάτι τέτοιο. Για μένα πιο χρήσιμο είναι να υπάρχει τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου και κατά την προετοιμασία και εκ των υστέρων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανωθούν οι εργασίες τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και η τελευταία μου πρόταση είναι να ξανασυζητήσουμε το θέμα σε ένα χρόνο όταν θα έχουμε συλλέξει κάποιες σχετικές εμπειρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σαλκαντράουι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο επί του περιεχομένου και θα επανέλθω στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να τον υπερτιμούμε, αλλά ούτε και να τον υποτιμούμε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Γιατί υπάρχουν κάποια θέματα αρκετά σημαντικά και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε το δικό μας ρόλο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση και τον όρο ότι μας αφορά το θέμα, μας ενδιαφέρει, είμαστε ενήμεροι και ε, όλα αυτά πριν επιτευχθεί μια συμφωνία. Εκ των υστέρων τι να το κάνεις, είναι δύσκολο να διαφωνήσεις. Ε, και αν το κάνεις έχει να κάνει με τη διαδικασία αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να ε, μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το βλέπει και να μας ενημερώνει τον των προτέρων για να μπορούμε σωστά να διαδραματίζουμε το ρόλο μας. Και λυπάμαι λίγο που ακόμα σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ανοίξει τα χαρτιά της. Γιατί εντάξει είναι γνωστό αυτό και σωστό για τη συμφωνία πλαίσιο ότι είναι έτοιμη, αλλά περίπου ένα χρόνο τώρα έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. Έτσι, θα πρέπει λίγο αυτό να μα προβληματίσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε σιγά σιγά ε, θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο, από ποια στιγμή και μετά. Παράδειγμα, όταν προτίθεται να ζητήσει μια εντολή από το Συμβούλιο ε, και όταν έρθει, ή μάλλον όταν έρθει η εντολή από το Συμβούλιο. Ποια ε, είναι η ώρα που μπαίνει και το Κοινοβούλιο στο παιχνίδι. Δεν θέλω να ισχυριστώ εγώ ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε συμφωνίες ξέρω εγώ, με τα νησιά Φίτζη αλλά όταν πρόκειται για συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Ρωσία που έτσι είναι και διαφορετική τάξη μεγέθους από τα Φίτζη υποθέτω ότι και στη διαπραγματευτική φάση ε, κάπου θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι και σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, να ενημερωνόμαστε, να μην μπορούμε να είμαστε και παρόντες, έτσι. Ε, αυτό ισχύει για πολλούς ενδιαφερομένους, όπως γίνεται στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί να είναι εκείνοι παρόντες ή όποιοι και εμείς να απουσιάζουμε. Εν πάση περιπτώσει, παρατήρηση αυτή, παρενθετικά, και περιμένω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από το Κοινοβούλιο, μεγαλύτερη σαφήνεια. Έρχομαι τώρα στο περιεχόμενο. Είχα την ευκαιρία το 2003 να συντάξω έκθεση για την ανάπτυξη μιας ατζέντα για την εξωτερική πολιτική ε, ε, μεταφορών και αεροπορικών και διαβάζοντας την έκθεση παραμένει επίκαιρη πρέπει να σας πω. Αυτό που μας ενδιαφέρει την είναι, να ανοίξει αγορά. Αλλά αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σύγκληση του ε, νομοθετικού περιεχομένου και του πλαισίου. Δηλαδή, εντάξει, να ανοίγει η αγορά ε, του ενός για τις εταιρείε του άλλου, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε περίπου και ίσους ε, κανόνες παιχνιδιού κάποια στιγμή. Και δεν έχω την εντύπωση ότι αυτό το έχουμε υπόψη μας και το αντιμετωπίζουμε με τρόπο συνεπή. Δηλαδή, εντάξει, να ρυθμίσουμε ε, τους κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά. Μετά τι γίνεται με τα κοινωνικά, με άλλα θέματα ασφαλείας, που και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ε, να μην υποτιμηθεί αυτό, να ε, πέσει σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό έχει να κάνει πούμε, τα δικαιώματα των επιβατών. Γνωρίζετε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, αεροπορικές ε, δεσμεύονται από κανόνε του παιχνιδιού που έχουμε ρίξει εμεί. Ξέρω εγώ, θυμάστε με την τέφρα ε, όταν ε, ξεράγει το ηφαίστειο έγιναν μεγάλες Και Οι Ευρωπαίοι πολίτες όμως που πετούσαν με άλλη εταιρεία, όχι η ευρωπαϊκή, δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα. Έτσι λοιπόν στο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τέτοιου στοιχεία στις ε, συμφωνίε για να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους οι πολίτες ανεξαρτήτω ε, εταιρεία από και προς την Ευρώπη. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι υπάρχει κίνδυνος τώρα για διάφορα παραθυράκια, γι' αυτό το τελευταίο, και πρέπει να το κοιτάξουμε οπωσδήποτε όταν συζητάμε για τέτοια θέματα ας πούμε, η πρόσβαση στο κεφάλαιο ε, αεροπορικών εταιρεών τρίτων χωρών. Πώς ρυθμίζεται αυτό. Εντάξει, κάνεις μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα και λες. Ανοίγουμε ένα στην αγορά στις εταιρείες του άλλου. Εκεί υπάρχει εκείνος κάποιοι τρίτοι που δεν έχουν καμία σχέση να αγοράζουν μερίδια των αεροπορικών εταιριών ε, με τις χωρών που έχουμε συμφωνίες εμείς και έτσι μπαίνουν από το παραθυράκι από την πίσω πόρτα και αυτοί στην Ευρώπη. Προσοχή όμως γι' αυτό, έτσι, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει και πάλι σε κατάχρηση των συμφωνιών αυτών από κάποιους τρίτους, ε, ε, κεφάλαια, διείσδυση άλλων κρατών, άλλων εταιριών, με τις οποίες όμως ακόμα εμείς δεν έχουμε συμφωνία. Έτσι. Και αυτό νομίζω δεν έχει ρυθμιστεί επαρκώς ή δεν, δεν το έχουμε σκεφτεί ε, επαρκώς. Ε, σταματώ εδώ, θέλω να ακούσω και τα δικά σα σχόλια και από πλευρά μου σίγουρα θα κάνω και προτάσεις για να βελτιώσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο για την δουλειά του. Είναι, είναι εισηγητής ε, στο όνομα όλων μας. Ε, έχουμε τώρα περισσότερα δικαιώματα από πριν, αλλά δεν είναι και τόσο παλά τη στιγμή που μπορούμε μόνο να πούμε ναι ή όχι. Και γενικά έχουμε περισσότερα δικαιώματα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά τα δικαιώματα πάντα συνδέονται με υποχρεώσει. Ε, γι' αυτό ε, δεν θα πρέπει ε, ελαφρά την καρδία να το πάρουμε το θέμα. Ε, από τη μία έχουμε κάποιε δυνατότητε, ο εισηγητή τι εξετάζει πιο προσεκτικά. συχνά λοιπόν λέμε πολύ βιαστικά ναι και θα πρέπει να προσέξουμε να μην πέσουμε στην παγίδα και ακριβώς αυτός είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε και φυσικά είναι καλό να υπάρχουν ε, συμφωνίες ε, με διεθνείς ε, αεροπορικές συμφωνίες αλλά και εδώ έχουμε πολλές ευθύνες και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Σκέφτομαι και αυτό που είπε ο Σάιντ Ελ Καντράουι όχι μόνο ε, για τις μεγάλες χώρες, ε, θα ήθελα και για τις μικρές ε, να γνωρίζω τι συμβαίνει. Και όπως είπε ο Μπράιαν Σίμψον, το όχι μπορεί να είναι θετικό, μπορεί, όπως στην περίπτωση SWIFT, μπορεί να δηλώσουμε έτσι μια πολύ ισχυρή θέση. Θέλουμε να έχουμε ε, καλά πρότυπα ασφαλείας. Ε, το θέμα όμως που τίθεται είναι τι γίνεται με την ανταλλαγή δεδομένων των επιβατών. Αυτό είναι ένα θέμα, πρόβλημα που έχουμε με τις ΗΠΑ ε, με το οποίο ασχολείται και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά τα δεδομένα των επιβατών σε αυτές τις ε, αεροπορικές ε, συμφωνίες ε, χωρίς να το γνωρίζουμε. Φυσικά, στις ε, διεθνείς ε, αυτές συμφωνίες. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια πρότυπα εντός και εκτός Ευρώπης. Δεν μπορούμε να επεκτείνουμε την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τι είναι σημαντικό για μας στις αεροπορικές μεταφορές και τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λίχτενπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν εμβαθύνουμε στο θέμα θα πρέπει να έχουμε κατά νου τι σκοπό έχουν όλα αυτά όσον αφορά την συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Ε, και εγώ συμμετείχα στην ε, συνέλευση και ήταν ε, σημαντικό με την εμπλοκή των των ε, προσώπων ε, του, λαού να ε, έχουμε πιο δημοκρατικές αποφάσεις. Σε μια τέτοια λογική λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουμε από νωρίς στις διαπραγματεύσεις ώστε να μην καταλήγουμε απλά σε ένα όχι και αυτό για μένα είναι αποφασιστικής σημασίας. Ελπίζω κανείς να μην αμφισβητεί ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ευρωβουλευτές ακόμα και αν κάποιοι από εμά δεν είναι κατά 100% προετοιμασμένοι και διατεθειμένοι να αναλάβουν το ε, σημαντικό αυτό έργο. Το θέμα όμως είναι πώς θα το κάνουμε ώστε να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Και ε, ο καλύτερος τρόπος εδώ είναι η ε, νωρίτερη ενημέρωση και η ε, συμβολή του Κοινοβουλίου πραγματικά να ληφθεί υπόψη και όχι απλά να μας παραμερίζουν και να μας λένε ότι α, δεν ξέρουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, τίποτα κοινοβουλευτικές ανοησίες είναι αυτές. Ε, ξέρω τις συζητήσεις αυτές ε, με έχουν ενημερώσει οι άνθρωποι που ξέρουν πώς λειτουργούν τα πράγματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα. Η συμβολή μας, ε, εάν θέλουμε να έχουμε την αποδοχή ε, του λαού, θα πρέπει να είναι πιο διαφανής και δεν θα πρέπει να καταλήγουμε σε διαμάχη μεταξύ διαφόρων ομάδων ενδιαφερόντων, διαφόρων λόμπι. Θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε κατά νου το στόχο αυτό και τότε θα είναι πιο σαφές πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να βρούμε μία στρατηγική ώστε η συμβολή του Κοινοβουλίου και ε, οι συνάδελφοι ήδη έχουν αναφέρει ποια είναι τα θέματα, είναι η προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, Αυτά είναι τα θέματα τα οποία μπορούμε ε, να επηρεάσουμε πετυχαίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε και θα πρέπει η συμβολή μας ε, να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ε, και όχι όπως στο παρελθόν που έχει αγνοηθεί η συμβολή του Κοινοβουλίου. Δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε, να, θέσουμε, να δημιουργήσουμε σωστές στρατηγικές, ε, να φροντίσουμε η συμβολή μας να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ώστε να μην καταλήγουμε απλά σε ένα διστακτικό ναι ε, με πολλές επιφυλάξεις ε, ή σε έναν όχι, ε, παραβλέποντας έτσι τα, τις θετικές πλευρές μιας συμφωνίας. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο ε, το εάν θα κάνουμε κάτι, αλλά και το πώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που εξηγήσατε τόσο καλά τις αλλαγές που έχει επιφέρει η συνθήκη της Λισαβόνα. Θα προσπαθήσω να τα πω απλά. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συμφωνία για τις υπηρεσίες οι οποίες υφίστανται εδώ και αρκετό καιρό. Και υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες που υφίστανται. Αυτό πρέπει, το είναι το πρώτο πρέπει να έχουμε κατά νου. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι και να αρχίσουμε να επαναδιαπραγματευόμαστε πράγματα που έχουν ήδη γίνει. Αυτό που ετέθη από πολλούς συναδέλφους είναι μια διαφορετική συμφωνία. Η συμφωνία για τους ανοιχτούς ουρανούς η οποία υφίσταται ακόμη και όπως λένε θα είναι η διαπραγμάτευση που γίνονται οι μεγάλες ε, διαπραγματεύσεις που παίζουν οι, μεγάλες, ε, οι μεγάλοι παίκτες. Νομίζω ότι θα πρέπει να την ελέγξουμε αυτή τη συμφωνία. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ομέρες Πολιτείες. Υπάρχουν τώρα άλλε ε, συμφωνίες υπηρεσιών που είναι υποδιαπραγμάτευση και οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει κάποια στιγμή κάπου να καταλήξουν. Κατά την άποψή μου, στο κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχει αλλάξει ο κόσμος γιατί έχουμε τη Συμφωνία της Λισαβόνας αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είμαστε εμεί οι διαπραγματευτέ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορεί που κάνουν ακριβώ αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ενημερωνόμαστε ή ότι δεν θα πρέπει να έχουμε εμπλοκή. Θα πρέπει όμω να γίνεται σε ένα επίπεδο πολύ ρεαλιστικό. Δεν θέλω να πω ότι η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να ελπίζω να μην φτάσει η Επιτροπή σε ένα σημείο όπου θα υπάρξουν μερικοί που θέλουν να πολιτικοποιήσουν μια τέτοια συμφωνία και ενδεχομένω έχουν το δικαίωμα του χρονοδιάγραμμα και θεωρούν ότι είναι το πλέον κατάλληλο μέρο για να θέσουν αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν... Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μίλησε πέντε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ηρέμησε για να μπορέσουμε να πούμε την άποψή μα. Ναι, εάν θε να μιλήσει, μπορεί να απευθυνθεί ε, στο Κοινοβούλιο. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Όπως έλεγα, Λοιπόν, δεν θα πρέπει να πολιτικοποιήσουμε τα όσα συμβαίνουν. Το θέμα είναι να έχουμε μία εμπλοκή. Εάν υπάρχουν συμφωνίες, είναι ε, σημαντικό εμείς στην Επιτροπή να μπορούμε να έχουμε κάποια άποψη. Όπως είπα, δεν θέλουμε έναν εμπορικό πόλεμο με καμία χώρα δεν έχουμε δικαιοδεσία σε τρίτε χώρε, σε πολλού τομεί. Σα είμαστε ρεαλιστέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Κύριε Πρόεδρε, είμαι σίγουρο ότι θα καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη προσέγγιση, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να είναι μια συζήτηση μεταξύ ενηλίκων. Ορισμένα πράγματα, για ορισμένα έχουμε ήδη αποφασίσει, άλλα θα αποφασίσουμε αργότερα. Και έχω τη βεβαιότητα ότι η Επιτροπή πει θα συμπεριλάβει αυτό το θέμα όπως πρέπει και ότι η Προεδρία θα υποβάλει μια ρεαλιστική πρόταση που μας βρει και εμάς συμφωνού. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ράνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα είπαν οι περισσότεροι, θα είμαι σύντομη, θα περιοριστώ σε μερικές παρατηρήσεις, μία ή δύο μόνο. Σε τέτοιου είδους συμφωνίες ε, η ε, στάση του Κοινοβουλίου και η ε, παρέμβαση του είναι το επισκεπτήριό του. Είμαστε οι μόνοι εκλεγμένοι και είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε να αποδείξουμε πόσο σοβαρά παίρνουμε τα μελήματα των Ευρωπαίων πολιτών που στο κάτω-κάτω μας εξέλεξαν εδώ. Και ως προς τις συμφωνίες που ισχύουν ήδη θα μπορούσαμε με ηρεμία, χωρίς να αναστατωθούμε, να ε, κάνουμε μια απογραφή, να διαπιστώσουμε ποια είναι τα προβλήματα, γιατί δεν έχουν λήξει ορισμένες συμφωνίες, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες, πώς πηγαίνουν. Και το ξέρω ότι στο τέλος μπορούμε να πούμε ναι ή όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε και συστάσεις φυλαχθούμε να μην κάνουμε τεχνικές υποδείξει. Στο κάτω-κάτω ούτε λόγος μας πέφτει γι' αυτό, ούτε είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Αλλά ε, είτε είναι μεγάλες ή μικρές χώρες ε, και δεν είναι μόνο η γεωγραφία, είναι και η οικονομία και πολλά τα στοιχεία μπορούμε να ε, συνεισφέρουμε και είναι και καθήκον μας εκτός από δικαίωμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να φερθώ σε ένα ή δύο σημεία. Όπως είπαν ε, και άλλοι ομιλητές, ε, πολλά από τα θέματα συζητήθηκαν ήδη. Στα πλαίσια της έκθεσης που θα πρέπει να κάνετε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι αυτές οι συμφωνίες είναι η κορυφή του παγόβουνου γιατί σύμφωνα με τη συνδίκη της Λισαβόνας έχουμε πολύ ευρύτερη ευθύνη για πολλές από τις διάφορες συμφωνίες που διαπραγματε... Ε, ε, τις διαπραγματεύονται σε όλους τους τομείς του εμπορίου. Νομίζω λοιπόν ότι η δική μου συμβολή είναι ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό στα πλαίσια ενός ευρύτερου θέματος που αφορά το νέο ρόλο του Κοινοβουλίου μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το δεύτερο σημείο είναι το εξή. Θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά το σχόλιο που έγινε από την Επιτροπή, ότι πραγματικά ελπίζω η Επιτροπή να δείξει κάποιο σοβαρότητα όταν λέει ότι θα εμπλακεί το Κοινοβούλιο. Οι παρατηρήσει που άκουσα δεν με κάνουν να νιώθω και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, ιδιαίτερη σιγουριά. Νομίζω ότι, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι άμεση, ντόμπρι, να μην παίζουν παιχνίδια. Γιατί εγώ τουλάχιστον θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όχι μόνο σε αυτή την επιτροπή αλλά και σε άλλες επιτροπές έτσι ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι υπάρχει αυξημένη δυνατότητα ελέγχου του Κοινοβουλίου. Πρέπει να έχουμε άμεση εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να ενημερωνόμαστε από την αρχή σε ό,τι αφορά την πορεία αυτών των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει συγκεκριμένη γνώμη όταν πρέπει να αποφασίσει ναι ή όχι στο τέλος. Και λέω σοβαρά στην Επιτροπή ότι εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτού του είδους τον απλό τρόπο ε, επικοινωνίας του Κοινοβούλιο θα, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με προβλήματα. Και γι' αυτό θα φταίτε εσεί. Παρακαλώ θερμά λοιπόν όταν θα έχουμε να κάνουμε με αυτά τα θέματα και σε αυτή την Επιτροπή και σε άλλε επιτροπέ, χρειάζεται λίγο περισσότερη εξέταση και για να διευκολυνθεί αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ανοιχτή και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη Επιτροπή και σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Μπράντμπερι. Αν θα μπορούσα να απαντήσω σε ορισμένα από τα θέματα που θίξατε, δίχως άλλο θα προσπαθήσω να Υποβάλλω μια εξισορροπημένη άποψη. Ο κύριος Μπραντμπορ και η κυρία Λούκτεμπερα έκαναν ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά την Επιτροπή. Μέσω της Γραμματείας προτείναμε η Επιτροπή να παρουσιάσει τα είδη των συμφωνιών και τα ωφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν στην τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά τι συμφωνίες με μερικές τρίτες χώρες. Η απάντηση ήταν ότι το, το έκαναν ήδη από το Μάρτιο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Παρόλα αυτά, όμως, μερικοί από εμά ε, δεν θυμόμαστε τι ακριβώς ε, ε, διεμήφθη το Μάρτιο. Θα ήταν λοιπόν μια καλή ιδέα να γίνει αυτή η εισαγωγική παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά τις εντολές, τα πρέπει να διερευνήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Επιτροπή. Από ό,τι φαίνεται εξετάστηκαν και συμφωνήθηκε ότι θα μπορούσαν να δοθούν οι εντολές σε εμπιστευτική βάση. Παρόλο που το πλαίσιο, η Συμβουλία πλαίσιο του 2005 και του 2010 δεσμεύονται, βάσει αυτό το συμφωνείο ε, δεσμεύονται να το κάνουν. Η Επιτροπή λέει ότι το εντολή είναι έγγραφο του Συμβουλίου. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να ξέραμε τι είναι αυτή η εντολή. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει ε, μέσα σε πλαίσια εμπιστευτικότητας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που αναζητάμε είναι λίγο περισσότερο πνεύμα συνεργασίας. Και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το εξετάσω λίγο περαιτέρω με την Επιτροπή. Κυρία Γέγκερ, θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο και να πείτε κάτι εξ ονόματος της Επιτροπής. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να τονίσω και πάλι ότι η Κομισιόν εμένει στην υποχρέωσή της να ενημερώνει άμεσα και πλήρως το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και κατά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Η Κομισιόν ενημερώνει το Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με την πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων προς το Συμβούλιο. Ε, επαναλαμβάνω, θα ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας άμεσα και πλήρως. Ε, γνωρίζουμε και τις ε, ρήτρες σχετικά με την προστασία της εμπιστευτικότητας. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο θέμα των αεροπορικών συμφωνιών. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω και αυτό. Εσείς ο ίδιος κύριε Πρόεδρε Αναφέρατε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις ε, διαπραγματευτικές ε, οδηγίες. Ε, θα πρέπει λοιπόν στην περίπτωση αυτή το Κοινοβούλιο να στρέφεται προς το Συμβούλιο. Ο κύριος Καντράουι ανέφερε το θέμα της συμμετοχής όπως και ο κύριος Μπράτμπορν. Οι αρμοδιότητες της Κομισιόν περιορίζονται ε, σε διεθνείς ε, διασκέψεις ε, και σε πολυμερείς συμφωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να το τονίσω αυτό και επίσης όλα αυτά υπόκεινται στις, στις διπλωματικές και άλλες δυνατότητες. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι πάντα ενημερώναμε την Επιτροπή σας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αεροπορικές συμφωνίες και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο από την ε, Διεύθυνση Ε που μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και θα ήθελα να επαναλάβω την ε, δέσμευση της ε, Κομισιόν να σας ενημερώνει άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά την προετοιμασία αυτών των συμφωνιών έχουμε μία, ένα καλό παρελθόν συνεργασίας με την Επιτροπή σας. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που έχουμε είναι η συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ξέρω ότι συνέβη με το Κοινοβούλιο, συνέβη και με εμά. Το γεγονό ότι μα λείπει ότι η δεύτερη φάση τη συμφωνία δεν πήγε τόσο μακριά όσο θα επιθυμούσαμε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πνευματικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα που δεν μας αναγνωρίζουν οι Αμερικανοί φίλοι δεν τα αγορίζουν ούτε και στους υπεύθυνους. Όπως γνωρίζετε σε ό,τι αφορά τα ιδιοκτησιακά αυτά ε, δικαιώματα, η καλύτερη συμφωνία ήταν αυτή που έγινε με τους Αμερικανούς φίλους. Ο κύριος Σαρκαντρά έκανε αναφορά πολύ σωστά στη ρυθμιστική σύγκληση. Θα ήθελα να πω για μία ακόμα φορά, το είπα και το Μάρτιο, το ξαναλέω και σήμερα, ότι για μας, στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών, των γενικών συμφωνιών, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρχει άνοιγμα της αγοράς χωρίς παράλληλα να υπάρχει ρυθμιστική σύγκληση. Γιατί, Γιατί αυτό σημαίνει συνθήκες για ε, ίσο ανταγωνισμό. Σημαίνει ικανότητα χρήσης των νέων δικαιωμάτων κυκλοφορίας ε, γιατί δεν θα είναι οι αρμόδιοι αντιμέτωποι με ασύμβατες, ασύμβατους κανονισμούς ή με μια υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτό που αναμένουμε από τη σύγκληση αυτή, αυτό είναι ένα θέμα που ε, υπάρχει σε όλες τις συμφωνίες και για ένα θέμα στο οποίο αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια των μεικτών επιτροπών που εφαρμόζουν αυτές τις συμφωνίες. Τι λοιπόν είναι η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών συμφωνιών σε σχέση με τις διμερείς συμφωνίες που κάνουν οι χώρες με ε, σε ατομική φάση με ε, τρίτες χώρες και που δεν έχουν διατάξει ε, για θέματα ε, σύγκλησης. Είτε αφορούν θέματα ασφάλειας, ανταγωνισμού. Δεν, δεν γίνεται όμως αναφορά σε δικαιώματα κυκλοφορίας. Αυτή η ισορροπία ε, είναι που θέλουμε να προωθήσουμε υπέρ των εμπλεκομένων αλλά και για να βελτιώσουμε το επίπεδο που δεν είναι πάντοτε το ίδιο παντού. Αυτή λοιπόν ε, η σύγκληση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσα από τις κοινωτικές συμφωνίες και όχι μέσα από τις διμερείς. Δύο τελευταία λόγια. Ο κύριος Μπρος έκανε αναφορά σε μία τακτική ενημέρωση. Ξέρετε ότι αυτό το συνέβη πριν από την ε, συμφωνία πλαίσιο. Θα συμβεί και με αυτή τη συμφωνία πλαίσιο η οποία υπεγράφει την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεσης προβλέπεται για την 31η Νοεμβρίου αρχές Δεκεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. 24-26 Ιανουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή, Μάρτιο 2011 ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Λοιπόν, χρόνο έχετε για να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα στη συζήτηση αυτή. Περιμέναμε τον πρόεδρο, τον ενδιαφέρει πρόεδρο στις 16 και 20 θα ήθελα να καλωσορίσω ένα πλόη συναδελφό μας, τον κύριο Βλόης Βάζεμπερκα. Θα θυμάστε ότι ο Φλόρες ήταν ένα ιδιαίτερο ενεργό μέρος της ομάδας των φιλελευθέρων για πολλά χρόνια. Mm. Φλόρες, ειλικρινά σε καλωσορίζουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ μου χρειάστηκε βέβαια κάποιο χρόνο, αλλά τα κατάφερα να φτάσω σε αυτή τη θέση. Ωραία. Τώρα, έχουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτών. Θερμή παράκληση μην να απομακρύνεστε, έτσι ώστε όταν φτάσει ο κύριος Σουτ να υπάρχουν και μερικά μέλη παρόντα για να μπορούν να του θέσουν ερωτήσεις. Τέσσερις και τέταρτο να είμαστε πίσω γιατί για πολλούς από εσά και τέταρτο θα γίνει και 20. Ευχαριστώ πολύ. If I could ask the contingent from the Kingdom of Belgium if they'd like to... Παρακαλώ τους πολίτες ε, του Βασιλείου του Βελγίου να καθίσουν καμιά ώρα να παλουκωθούν να ακούσουν τον Υπουργό τους. So, ladies and gentlemen, it's... Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα να σας παρουσιάσω τον Υπουργό Σουτ, Σουτ ο οποίος θα προβεί σε μία αξιολόγηση του πρώτου εξάμεινου της Βελγικής Προεδρίας. Και θα μας μιλήσει για την ε, συνάντηση του Συμβουλίου. Κύριε Γραμματέ, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Μπράιαν. Αγαπητοί συντονιστέ. Α, βάλτε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω Ολλανδικά. Αγαπητοί συντονιστές, εισηγητές, καθώς και μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτής της ανταλλαγής απόψεων με πολύ μεγάλη χαρά θα σας ενημερώσω για την κατάσταση των πραγμάτων και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, καθώς επίσης και τις δράσεις που αναμένονται στο πρόγραμμα προτεραιοτήτων, το οποίο σας παρουσίασα στις 13 ε, Ιουλίου ενεστώτος έτους. Στο μεταξύ θα γνωρίζετε χωρίς καμία αφιβολία ότι το βιώσιμο μέλλον των μεταφορών καθώς επίσης και ασφάλεια ε, ενεργητική και επαθητική για όλα τα μέσα μεταφοράς είναι λέξεις κλειδιά για το πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας και είναι και πρόκληση μεγάλη για το μέλλον των μεταφορών. Πρώτη μας προτεραιότητα στην αρχή της Βελγικής Προεδρίας ήταν η παρουσίαση της Λευκής Βίβλου για το μέλλον των μεταφορών. Ποιες απαντήσεις θα πρέπει να δώσουμε στις νέες προκλήσεις για τις μεταφορές. Να δούμε πώς ε, μπορούμε να εγγυηθούμε τον ε, ίσο ε, ανταγωνισμό όλων των μέσων μεταφορών. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε, μάλλον ε, ανακοίνωσε ότι θα φτάσει η Λευκή Βίβλος ε, το 2011 μόλις, παρόλο που τα θέματα επήγουν. Δεν θελήσαμε λοιπόν εμείς να περιμένουμε με αδράνεια την άφηξη της Λευκής Βίβλου. Κατά τη διάρκεια του ε, προηγουμένου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών ακριβώς διοργανώθηκε μια αλλαγή απόψεων για αυτή τη Λευκή Βίβλο με δύο συγκεκριμένα ερωτήματα θελήσαμε από το Συμβούλιο να δώσουμε την απαραίτητη υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την κατάρτιση της Λευκής Βίβλου. Και τα δύο ερωτήματα ήταν τα εξής. Πρώτον, ποιες πρέπει να είναι οι γενικές προτεραιότητες και απαντήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφορών για την επόμενη δεκαετία θέλουμε να αγγιθούμε μια βιώσιμη και υφόρο ανάπτυξη στις μεταφορές και να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις, είτε πρόκειται για προβλήματα περιβαλλοντικά, την κλιματική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση ή τη γύραση του πληθυσμού, ε, τις μεταναστεύσεις, ε, την εξάντληση ορυκτών ε, πόρων, αστιφιλία, εξωτερήκευση του εξωτερικού κόστους και ε, ε, ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων μέσων μεταφορών. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση ε, έχει ως εξής. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε η ανάπτυξη και η χρήση των νέων τεχνολογιών να μπορούν να διαδραματίσουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία ενός βιώσιμου και ε, σωστού συστήματος μεταφορών μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και να εγγυηθούν ε, την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και μάλιστα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και την οικονομία και ταυτόχρονα να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και να αυξάνουν την ασφάλεια των μεταφορών. Πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι η θέση των νέων κρατών μελών Ε, είναι κάτι το οποίο ε, μας ε, προβληματίζει. Ορισμένα κράτη θέλουν μεγαλύτερες υποδομές, περισσότερο εξυγχρονισμό. Άλλα κράτη θέλουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Δηλαδή είναι ευρύ ε, το ε, επίπεδο. Ο Επίτροπος Κάλλας ζήτησε συγγνώμη πρέπει να σας πω για την καθυστέρηση της Λευκής ε, Βίβλου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυτής. Κατά τη διάρκεια του ίδιου Συμβουλίου παρουσιάστηκε μια πρόταση οδηγίας για την αναδιατύπωση του πακέτου Recast, ε, του πρώτου πακέτου των σιδηροδρόμων. Για τις χερσαίες μεταφορές και την ομάδα εργασίας γνωρίζετε ότι η ομάδα αυτή στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών θα ε, παρουσιάσει μια έκθεση και η επόμενη Προεδρία που είναι Ουγγρική έχει ε, θέσει το θέμα αυτό ως προτεραιότητα. Τους περασμένους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίση το τέταρτο πρόγραμμα δράση για την ασφάλεια των μεταφορών. Στι 2 Δεκεμβρίου ε, θέλουμε να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο προ έγκριση τα συμπεράσματα αυτή τη προσπάθεια. Ε, ε, στη συνέχεια μπορώ να σας πω ότι στο θέμα της διασυνοριακής κυκλοφορίας και επιβολής του νόμου έχει γίνει μεγάλη πρόοδος προς μια συνένεση και στόχος είναι να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στις 2 Δεκεμβρίου, όπως σας είπα και προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι, οι προσδοκίες ε, από τις διαπραγματεύσεις που τρέχουν τα δικαιώματα για τους επιβάτες των λεωφορείων είναι δύσκολο όμως να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα. Έχουμε σε κάθε περίπτωση δεσμευτεί να καταλήξουμε σε μια ρύθμιση, σε μια συμφωνία εφαρμόσιμη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι ακόμα σε θέση ειλικρινά να σας πω προς τα πού προσανατολίζεται αυτή η πρόταση. Πρόεδρε, είμαι πεπισμένος ότι η μεγάλη κινητικότητα ε, αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνοδεύεται με τη μέγιστη ε, μέρημνα για το περιβάλλον. Επίσης να βελτιστοποιηθούν όλοι οι τρόποι μεταφορών, όλα τα μέσα μεταφορών με τρόπο πιο οικολογικό και πιο καθαρό. Διόδια. Και, ε, που να εξαρτώνται από την απόσταση που διανύεται, από το χρόνο ε, χρησιμοποίησης ε, ε κάποιων ε, δρόμων και εσωτερική συγγνώμη του εξωτερικού κόστους είναι μερικά μόνο ε, στοιχεία και πτυχές. Και μπορώ να σας δηλώσω έτσι και με κάποια περηφάνεια ότι ε, στο περασμένο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών επιτέλους επιτύχαμε μια πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση της Ευρωβινιέτας. Υποθέτω ότι στο μεταξύ έχετε ενημερωθεί σχετικά και εσείς. Παρ' αυτά επιτρέψτε μου να σας επαναλάβω τα σημαντικότερα έτσι, σημεία για κάθε σαφήνεια. Έχουμε μια βάση τώρα για την αναθεώρηση που επιτρέπει ότι το εξωτερικό κόστος όπως είναι η ρήπανση της ατμόσφαιρας και η χορύπανση ε, εσωτερικεύονται με βάση τα διάφορα πρότυπα Euro, Euro 0, 1, 2, 3, 4, τα γνωρίζετε, σύμφωνα με την αρχή ότι ο ρηπαίνων πληρώνει και ο ρηπαίνων περισσότερο πληρώνει περισσότερο. Επίσης, έχουμε και μια ισόρροπη λύση για την κυκλοφοριακή συμφόρηση ε, με προσαρμογή του τέλους κυκλοφορίας ε, για τις υποδομές και ένα κόστος που μπορεί να φτάνει μέχρι το 175% ε, του αρχικού διοδίου σε 5 ώρες εχμής. Έτσι θέλουμε με υψηλότερα διόδια, με ε, υψηλότερα τέλη κυκλοφορίας να αποθαρρύνουμε τους οδηγούς φορτηγών να χρησιμοποιούν τους δρόμους κατά τη διάρκεια των ωρών εχμής. Έτσι το τελικό κόστος είναι ουδέτερο και τι σημαίνει αυτό ε, να έχουμε και αντίστοιχη μείωση σε σχέση με το βασικό τέλος κυκλοφορίας στις ε, ε, λεγόμενες νεκρές ώρες ή ώρες που η κυκλοφορία είναι πολύ λιγότερη από τις ώρες εχμής. Προβλέπονται επίσης και κάποιες εξαιρέσεις χρονικές για οχήματα τύπου Euro 5 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010 και του 2017 για το Euro 6. Ελαφρύς λοιπόν και εξαιρέσεις που σημαίνουν ενθάρρυνση ακριβώς ε, για τη χρήση ε, οχημάτων που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και είναι πιο φιλικά. Άλλο βήμα, πιο ε, αϊφόρες μεταφορές, πιο πράσινες μεταφορές και σύνδεση της ακτοπλοείας με τις εσωτερικές ναυσιπλοείας. Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, ε, είχαμε ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργομεταφορών στην Αμβέρσα για τη μεταφορά ε, από τη θάλασσα στις εσωτερικές πλωτές οδούς με αρμόδιους φορείς. Blue Belt και Blue Lane ε, λέγονται αυτά τα συστήματα για μεγαλύτερη ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου ε, ναυσιπλοείας. Αυτό τα έχει περιγράψει σε αδρές γραμμές ήδη από πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον η, η έμσα, συγγνώμη, η ε, αρμόδια υπηρεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα θα κάνει προτάσεις ε, και η ομάδα εργασίας που επιφορτίζεται ε, με αυτά τα θέματα θα κάνει πρόταση στο Συμβούλιο, μάλιστα στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών. Επίσης, περιμένουμε να δημοσιευθεί η πρόταση της ΕΜΣΑ ε, ως προς την αναθεώρηση του ρόλου και της αρμοδιότητας της ναυτιλιακής υπηρεσίας στη Λισαβόνα που ρυθμίζεται ε, από τον κανονισμό 1406 του 2002. Η έγκριση του πακέτου ΕΡΙΚΑ 3 ε, περιλαμβάνει τις περισσότερες από αυτές τις αρμοδιότητες και εξουσίες. Κανονικά, στις 28 Οκτωβρίου αναμένεται η ε, έκθεση αυτή το πόρισμα έτσι ώστε στο επόμενο ε, Συμβόλιο να παρουσιαστεί μόνο μια έκθεση πρόοδου. Σε κάθε περίπτωση το Βέλγιο θα ε, εξακολουθεί να πιέζει σε αυτό το θέμα ε, ακριβώς και βάσει των δεσμεύσεών μας για την ομάδα εργασίας για, τις, για την αυσιπλοεία και κατά τη διάρκεια, ξέρετε, της Ουγγρικής Προεδρίας θα διατηρεί το Βέλγιο την Προεδρία αυτής της ομάδας για τη θάλασσα και την αυσιπλοεία. έρχομαι τώρα στις αναέριες μεταφορές. 37η ε, ε, ε, συνεδρίαση του ΙΚΑΟ στο Μόντρεαλ. Που, ΙΚΑΟ που είναι ο Διεθνής Οργανισμός Αέριας Κυκλοφορίας. Τέλη Σεπτεμβρίου γνωρίζετε ότι διεξήχθη αυτή η συνεδρίαση, συμμετείχαμε κι εμείς και πρέπει να σας πω ότι μπορεί να είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα ως προς την ασφάλεια, την ενεργητική και παθητική αλλά και το περιβάλλον. Κυρίε και κύριοι, το σημαντικότερο αλλά και το δυσκολότερο ήταν οι σχέσεις μεταξύ της ε, διεθνούς ε, πολιτικής αεροπορίας και τι επιπτώσει που έχει στο κλίμα. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να υπογραμμίσω ότι η συμφωνία που επετέφθη ήταν ιστορική κατά την άποψή μου. Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, η Γενική Συνέλευση του ΙΚΑΟ και ε, λόγω της πίεσης που δέχτηκα ε, από τα ευρωπαϊκά κράτη και το λόμπι κατέληξε σε ένα ψήφισμα για τον περιορισμό ε, των ενετικών συνεπειών της ενέργειας κυκλοφορίας στην κλιματική αλλαγή. Με ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα είναι ο ηρμός για τα κράτη-μέλη του ΙΚΑΟ που είναι 190 για τα επόμενα 40 έτη. Συνεπώς, στα ε, πλαίσια και στον τομέα της εναέρειας κυκλοφορίας μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κυρίες και κύριοι, ε, και να σας ανακοινώσω ότι ε, το μεσημέρι κήρυξα την έναρξη μιας ημερίδας, μάλιστα δύο ημερών, στην Μπρουζ για τα θέματα αυτά, για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πολιτικής αεροπορίας, η ασφάλεια ενεργητική και απαθητική της αέρας κυκλοφορίας, ε, το ΣΥΣ2 και την κλιματική αλλαγή. Οι ενδιαφερόμενοι ε, που συμμετέχουν πάνω από 350 από όλα τα κράτη είναι παρόντες στη σύνοδο αυτή κορυφή στην Προύζ. Στόχος ποιος είναι. Οι συζητήσεις εκεί ε, να ε, ε, καταλήξουν σε μια διακήρυξη για αυτά τα θέματα, η λεγόμενη διακήρυξη της Μπρουζ για την πολιτική αεροπορία, για την εναέρεια κυκλοφορία. Και τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι σε συνεργασία με το τρίο την Ισπανία και την Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, συμφωνήσαμε για το μέλλον της ε, υπηρεσίας GNSS για το σύστημα πλοήγησης ε, ε, ως προς τα θέματα ασφαλείας και διαπίστευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει και καλύτερα στις ενέργειες εκεί ε, και ο κανονισμός 19-12 του 2010 δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου και θα τεθεί σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου. Στις 24 Ιουνίου του 2010 κατέθεσε ένα πρόγραμμα δράσης η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για το GNSS και αυτό εγκρίθηκε. Ο κανονισμός 683 του 2008 ε, αναφέρεται σε μια διάμεση αναθέωση του 2010 για τον τρόπο διαχείρισης του συστήματος GNSS με την αντίστοιχη ανάλυση κινδύνου, τη διαχείριση και ανάθεση συμβάσεων στην ε, βιομηχανία, καθώς επίσης και την προβληματική χρηματοδότησης. Ακόμα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταθέσει αυτή την αναθεώρηση. Αυτά ε, συνοπτικά κύριε Πρόεδρε, τα πιο σημαντικά στους διάφορους κλάδους των μεταφορών για τους επόμενους μήνες. Ε, ελπίζω να μας βοηθήσει και στην προσπάθειά μας αυτή και το Κοινοβούλιο και είμαι στη διάθεσή σας για όποια ερώτηση θέλετε να μου κάνετε σχετικά. Okay, President in Office, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν τα πρακτικά. Μέχρι τώρα έχω τον κύριο Κρός, τον κύριο Αλκατράου, την κυρία Μάισνερ, Κράμερ, ε, Ζήλα από τους συντονιστές, την κυρία Τεβέιρακ, τον κύριο Λάχτφριντ, Λίχτανπεργκερ και άλλους ομιλητές. Υπάρχει άλλος που θέλει να πει στο κατάλογο. Πείτε το τώρα. Ίσο, πάστε για πάντα. Ωραία. Συντονιστές από τρία λεπτά. Οι υπόλοιποι βουλευτές δύο λεπτά, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. ο κύριος Κρός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Προεδρεύοντα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ε, την ενδιάμεση αναθεώρηση. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχετε προχωρήσει περισσότερο ε, στο μέσο της Προεδρίας σας από ότι άλλες Προεδρίες ε, στο τέλος τους. Ε, είναι ίσως λοιπόν αυτό ο καλός ιονός για θέματα που εκκρεμούν ακόμα για το μέλλον. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλά θέματα, αλλά αναφερθήκατε στην ασφάλεια και την βιωσιμότητα. Ε, έχετε προχωρήσει πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις αυτές και είναι σαφές ότι ήταν τολμηρό να θέσετε το θέμα της ευρωβινιέτας ε, στην ημερησία διάταξη. Αυτό το θέμα μπορεί να αποτελέσει επιτυχία για μας εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και κάποια ε, θέματα παραμένουν εκκρεμή. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την ε, αφοσίωσή σας ε, στο μη νομοθετικό τομέα. Σκέφτομαι την οδική ασφάλεια. Γιατί επειδή είναι πολύ σημαντικό και για μας το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο να ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά ώστε οι πολίτες να ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν τους πολίτες πολύ πιο πολύ από την νομοθετική δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα και ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ συγκεκριμένα βήματα προόδου, να μπορέσουμε να προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, να μην παραμείνουμε στην θεωρία. Ως προς αυτά που έχουν αποφασιστεί, είναι καλό το ότι έχετε ξεκινήσει τις συζητήσεις στο Συμβούλιο για τη Λευκή Βίβλο. Δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, έστω και με καθυστέρηση να παρουσιαστεί φέτος η Λευκή Βίβλος αυτή ε, και σε συνεργασία μαζί σας και κατόπιν με το Συμβούλιο να μπορέσουμε να θέσουμε τα σημαντικά θέματα. Αυτό θα πρέπει να γίνει πριν το 2011 πιστεύω. Ε, κάτι άλλο. Όταν ε, κοιτώ το θέμα της Ευρωβινιέτας, ε, όπως έχω πει, χαίρομαι πολύ με το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Ευρωβινιέτα έχει νόημα μόνο εάν συμμετέχουν όλοι. Αν συνεχίσει να αποτελεί εξαίρεση για κάποιους, τότε δεν θα έχει πολύ νόημα η εσωτερικεύση του κόστους. Επίσης, έχουν γίνει προσπάθειες να βρεθούν λύσεις, αλλά εάν ε, οι μεταφορές ε, εξυπηρετούν ε, στην βελτίωση της κινητικότητας, τότε Πράγματι έχουμε πετύχει, αλλά ε, δεν μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε κάθε τέσσερα χρόνια. Παρακαλώ να το μεταφέρετε αυτό στου συναδέλφου. Δεν μπορούμε κάθε πέντε χρόνια να υιοθετούμε ένα ωραίο πρόγραμμα. Ε, Όποιο ξεκινήσει πρέπει να δώσει και συνέχεια. Εάν ε, το ε, Α είναι ο προγραμματισμό, ε, εάν δεν φτάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η χρηματοδότηση, τότε δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Και επίση μια τελική παρατήρηση για τα δικαιώματα των επιβατών, κύριε Πρόεδρε Πρόεδρε, είσαστε ρεαλιστή υπουργό, αλλά πραγματικά εδώ στο Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμού και στο πεδίο εφαρμογή και στα δικαιώματα. Κάτι θα πρέπει να απομείνει ώστε να έχουμε κάποια αξιοπιστία ε, στου ανθρώπου ε, τη Ευρώπη. Σας ε, παρακαλώ λοιπόν να λάβετε υπόψη το αίτημά μου αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκρό. Ε, Συνήθω τηρείτε το χρόνο σας. Ε, σήμερα δεν ήσασταν τόσο καλό. Ο κύριο Αλκαντράου, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά εξ ονόματο της ομάδας μου θα ήθελα να πω ότι προς το παρόν είμαι ικανοποιημένο με τα όσα έχετε πράξει. Έχουμε όλη την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια πρόοδος τώρα σιγά σιγά στις εργασίες του Συμβουλίου και πάει καιρό που δεν είχαμε αυτή την αίσθηση. Πολύ θετικό είναι αυτό για εσά. Πλην όμω έχει σημασία όχι μόνο να συμφωνεί στο Συμβούλιο στους κόλπους του, αλλά τελικά να επιτευχθεί συνολική συμφωνία και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά θεμάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Βλέπε Ευρωβινιέτα, βλέπε δικαιώματα επιβατών, βλέπε διασυνοριακές ε, ε, ε παραβιάσεις ε, κυκλοφορία. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά και δεν είναι μόνο το κερασάκι στην τούρτα. Και εδώ και μήνες εκκρεμούν αυτά τα θέματα και έχουν αποτελματωθεί. Εκφράζω και εγώ τη θλίψη μου μαζί σας ότι δεν μπορεί να γίνει επίσημη ακόμα συζήτηση για τη Λευκή Βίβλο αλλά και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα. Συμπέρασμα, θα πρέπει να είναι το σύστημα μεταφορών μας και πιο αποτελεσματικό και πιο βιώσιμο και χρειάζεται εδώ ένα μείγμα ε, μέτρων και τιμολόγηση. Και έρχομαι στην ε, Ευρωβινιέτα. Το γεγονός ότι έχετε πετύχει η πολιτική συμφωνία από μόνο του είναι σημαντική είδηση. Γιατί Είχαμε αποθαρρυνθεί από το Μάρτιο του 2008 που στο Κοινοβούλιο πετύχαμε μια συμφωνία. Υπάρχουν όμως μεγάλες ε, διαφορές ακόμα για το κόστος, το εξωτερικό και πώς θα γίνει αυτό μεταβατικές ε, λύσεις, ε, κλήσεις, εξαιρέσεις και τα λοιπά προσωρινές. Θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Ελπίζω να γίνει αυτό κατά τη διάρκεια της δικής σας Προεδρίας, να δούμε μήπως μπορεί να υπάρξει κάποια προσέγγιση ε, και ελπίζω να δεσμευτείτε και για την ασφάλεια ε, στην ε, οδική κυκλοφορία και τις παραβάσεις στις διασυναριακές έχει γίνει μεγάλη φασαρία και διαπληκτισμό τελευταία για την νομική βάση αλλά το θέμα είναι οδική ασφάλεια και οι ζωέ των ανθρώπων κάποια στιγμή βρείτε τα εν πάση περιπτώσει για τις παραβάσεις στο ε, σύνολο και για τα δικαιώματα των επιβατών το τελευταίο βεβαίως είναι απαράδεκτο να αποδυναμωθεί τελείω μέχρι να μείνει καινογράμμα Δεν μπορούμε να το δεχθούμε και περιμένουμε από το Συμβούλιο κάποια ευελιξία να σκεφτεί πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογή και να δώσετε και κάποιο περιεχόμενο σε αυτά τα δικαιώματα. Συνοψίζω λέγοντα ότι Προς το παρόν, πώς να το πω, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε επιτυχημένη την Προεδρία σας, αλλά ελπίζουμε τους επόμενους δύο-τρεις μήνες ε, και στο τέλος να έχουμε την ευκαιρία να πούμε ότι ήταν εξαιρετική άριστη η Προεδρία, όχι μόνο ικανοποιητική. Υπάρχουν θέματα που δεν έχετε ακόμα αντιμετωπίσει, όπως ε, οι κανόνες παιχνιδιού για τη χρηματοδότηση μέσων ασφαλείας θα τα πει ο συνάδελφος αυτά, Λάιχτφριντ, κατά τα άλλα συνολικά θετικά τα βλέπω. Ευχαριστώ. Κυρία Μάισνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν χρειάζεται να επαναλάβω πολλά από όσα υπόθηκαν, οπότε μην ανησυχείτε, δεν θα ξεπεράσω το χρόνο μου. Ε, στην αρχή της Βελικής Προεδρίας υπήρχε ε, εν μέρη ο φόβος ότι ε, οι δυσκολίες ε, για την διαμόρφωση κυβέρνησης θα μπορούσαν να προκαλέσουν εμπόδια. Ε, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι αξιέπαινο από εσά το ότι προσπαθήσατε να προωθήσετε τα θέματα. Ε, η Κομισιόν έχει υποβάλει κάποια, ε, κάποιες προτάσεις, αλλά τα περισσότερα τα δούμε του χρόνου. Όσον αφορά την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ε, και το πακέτο των σιδηροδρόμων και θα, αυτά θα πρέπει να συζητηθούν. Δεν μπορείτε όμως να πετύχετε εδώ ε, λύσεις μέσα σε ένα εξάμεινο. Πολύ συγκεκριμένα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα. Πρώτον, τα δικαιώματα των επιβατών. Ο εισηγητής ε, μίλησε πολύ ε, έντονα, κάτι πρέπει να γίνει εδώ ε, και θα είναι αξία αν μπορείτε επί Βελγικής Προεδρίας να πετύχετε ε, καλά αποτελέσματα ως προς ε, τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ελπίζω να τα καταφέρετε. Ίσως καταφέρουμε πράγματι να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Όσον αφορά την Ευρωβινιέτα, όσον αφορά την πολιτική μεταφορών, είναι κρίμα το θέμα που έχει να κάνει με την δέσμευση των χρημάτων για συγκεκριμένους στόχους. Μόνο όταν ξέρει κανείς ε, τι χρειάζεται από χρήματα ε, στον τομέα των ε, μεταφορών και κατά πόσο πρέπει να μειώσει τις εκπομπές θα μπορέσει να καταλήξει σε καλά αποτελέσματα. Και επίσης όσον αφορά τις ολοκληρωμένες ναυτιλιακές μεταφορές είχα ήδη την πρώτη μου έκθεση και ε, για εσά του Βέλγου. Ε, αυτό αποτελεί σημαντικό θέμα. Ε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Όσον αφορά την αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων τη ΕΜΣΑ, έχουμε ήδη πει ότι θα πρέπει να εξεταστεί τι περαιτέρω αρμοδιότητε θα μπορέσει να έχει η ΕΜΣΑ ώστε να αποφευθούν καταστροφές από πετρελοκυλίτες στο μέλλον. Κάνετε λοιπόν πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ για το όσα έχετε πετύχει μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Παραμείνατε εντός του χρόνου. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και όπως ήδη υπόθηκε όταν ε, συγκρίνει κανείς τις διάφορες προεδρίες έχετε πετύχει πάρα πολλά ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυθείτε. Ε, και δεν είμαστε πάντα ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, είμαστε όμως απόλυτα ικανοποιημένοι με τη δουλειά σας. Ως Γερμανός ε, μπορώ να πω ότι προφανώς είναι καλύτερο το να ζει κανείς σε χώρα χωρίς κυβέρνηση παρά με μια αδύναμη κυβέρνηση. Ναι, όλοι ε, γελάνε, ε, πάση πτώση. Ε, γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Θα ξεκινήσω από την Ευρωβινιέτα. Το θέμα δεν είναι να πάρουμε χρήματα από τον τομέα των μεταφορών για να ε, ε, εξηγιάνουμε ε, την κρατική οικονομία. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Κάθε αυτοκίνητο στην Γερμανία επιδοτείται ε, με 3.000 ε, ευρώ ε, και το θέμα είναι αυτά τα χρήματα να επιστρέψουν στον προϋπολογισμό για να χρηματοδοτηθούν άλλοι τομείς. Πρόκειται λοιπόν για ένα μικρό βήμα. Έτσι πρέπει να αναγνωρίσουμε την εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους ε, αλλά ε, το κόστος για το κλίμα, για παράδειγμα, δεν έχει ληφθεί σχεδόν καθόλου υπόψη ε, και έχουν, έχει καταργηθεί εδώ το κόστος για την συμφόρηση. Είναι ένα μικρό βήμα, αλλά ελπίζω να καταφέρουμε περισσότερα, διότι συνεχίζουμε να έχουμε άδικη, άδικο ανταγωνισμό για ε, στις συντηρηδρομικές μεταφορές, για παράδειγμα, ε, δεν υπάρχει πλαφόν ε, στο συγκεκριμένο θέμα, σε αντίθεση με τι οδικές μεταφορές. Δεν θα μπορέσουμε... Ε, λοιπόν, να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος εάν ε, δεν λάβουμε υπόψη μας τις μεταφορές που ευθύνονται για το 30% των εκπομπών. Επίσης, όσον αφορά Επίσης έχετε προχωρήσει πάρα πολύ καλά όσον αφορά το θέμα των ε, φορτηγών κτλ. Η Ελβετία το έχει κάνει πολύ καλά αλλά δεν ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, ασφάλεια, η οδική ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ε, θέλουμε να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, έχουμε προτείνει να υπάρχουν όρια ταχύτητας εντός των πόλεων. αυτό θα βοηθήσει την αποδοχή και την οδική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ελέγχους φυσικά. Και το ίδιο ισχύει για την κατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχώς ε, είσαστε ο ο τρίτος ή τέταρτος ε, ε προεδρεύοντας που, δεν έχει αναφέρει ε, την σύμβαση των Άλπαιων και Επίση, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβετών, θέλουμε τα ίδια δικαιώματα για όλου. Δεν είναι δυνατόν ε, στο, στις μεταφορές να πληρώνεται αποζημίωση μετά από μία ώρα ενώ στις αεροπορικές μετά από τρεις ή πέντε ώρες. Ε, θέλουμε λοιπόν ε, τα ίδια δικαιώματα για όλους τους επιβάτες. Ε, και ε, θέλουμε λοιπόν ακόμα και για τους επιβάτες ε, λεωφορείων ε, τα ίδια δικαιώματα. Ο κύριος Ζήλερ, τελευταίος ομιλητής αυτόν τον γύρο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, την Προεδρία για την ενδιάμεση αυτή αναθεώρηση. Πιστεύουμε ότι έχετε πετύχει πολλά στον τομέα των μεταφορών. Πιστεύω ότι η δύσκολη πολιτική συμφωνία που αφορά την Ευρωβινιέτα που ε, υιοθετήθηκε με πολύ μικρή πλειοψηφία είναι σημαντικό επίτευγμα. Θα ήθελα να αναφερθώ όχι τόσο πολύ στα ε, δικαιώματα των επιβατών, διότι υποθέτω ότι ε, γνωρίζετε την έλλειψη ε, προόδου στι συγκεκριμένε διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στην ε, κατάσταση στον ε, τομέα των αερομεταφορών. Πιστεύω ότι στο Μοντρεάλ έχουμε δει πολύ θετικές εξελίξεις, ωστόσο οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ε, πολύ υψηλό κόστος για τις υπερτήσεις ε, τους στην Σιβηρία. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το θέμα αυτό. Τέσσερες χώρες έχουν διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία και δεν πληρώνουν τα τέλη αυτά. Βλέπετε να μπορεί να υπάρξει πρόοδος στο θέμα αυτό. Και κατά τη συνάντηση στην Μπρουζ θα μπορούσε να συζητηθεί αυτό ή ε, βλέπετε να υπάρχουν άλλα φόρουμ που να μπορεί ε, να ε, συζητηθεί το θέμα αυτό και όσον αφορά τις εκπομπές θείου που, αυτή τη στιγμή και την ε, σύμβαση Μαρπόλ. Ε, αυτή τη στιγμή ε, μόνο η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα καλύπτονται από τον περιορισμό για τι εκπομπέ θείου. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού, διότι κάποιε χώρε δεν δεσμεύονται από του κανόνε αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Προεδρεύοντα, θέλετε να απαντήσετε στου πέντε πρώτου ομιλητέ και κατόπιν να προχωρήσουμε στο δεύτερο γύρο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πρώτον, για την Ευρωβινιέτα. Να σας πω. Πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις περιφερειακές και τις κεντρικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τη γεωγραφική τους δηλαδή θέση. Είναι πάρα πολύ διαφορετικές οι θέσεις τους έτσι, και πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Οπότε, ε, πώς να το ονομάσω, ότι είναι τη μέθοδος της εξομολόγησης. <laughs> Για να ε, εκτιμήσουμε τις διάφορες θέσεις και τις ε, γενικές αρχές. Γιατί καμιά φορά όμορες χώρες που συνεργούν μεταξύ τους δηλαδή, στις Άλπεις για παράδειγμα, έχουν διαφορές. Δεν χρειάζεται να αναφέρω χώρες για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Ξέρουμε ότι εκεί οι ε, θέσεις ήταν ε, πολλές φορές αντικρώμενες λόγω και συμφερόντων. Και χρειάστηκε να βάλουν και οι δύο πλευρές νερό στο κρασί τους για να καταλήξουμε κάπου. Και χρειάστηκε πραγματικά να κάνουμε τάμα για να ε, τους φέρουμε στην ίδια θέση και τους δύο. Σε ό,τι αφορά την Ευρωβινιέτα, ως προς την αρχή την ίδια, συμφωνούσαμε και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο βαθμός ρήπανσης και να δοθούν και κίνητρα έτσι ώστε οι μεταφορές να είναι όσο πιο πολύ οικολογικές, όσο πιο οικολογικές γίνεται δηλαδή και φόρες στο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα, τα περιαστικά και διάφορους άξονες που ε, εμφανίζεται ε, συμφόρηση ή μπορεί να ε, έχουν κορεσμό. Και, λοιπόν, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις αρχές πρώτον και να λάβουμε όλη υπόψη ε, ότι υπάρχουν ενδεχομένω κάποιες λύσεις για ειδικά προβλήματα κάθε χώρας. Γνωρίζω δε πάρα πολύ καλά ότι η φόρμουλα, ο τύπος που επεξεργαστήκαμε είναι μια συμφωνία πλαίσιο τρόπον τεινά. Διότι έχουν οι διάφορες χώρες ακόμα ε, περιθώρια ελιγμών για να προσδιορίσουν ε, τι θα κάνουν. Πάντω είναι αναπόφευκτο κυρίε και κύριοι γιατί τα προβλήματα των διαφόρων χωρών διαφέρουν πάρα πολύ και είναι και στην πραγματικότητα πάρα πολύ διαφορετικά και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Ε, και θα πρέπει να μπουν μερικέ παράμετροι στην Ευρωβινιέτα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ειδικά προβλήματα, με ειδικά μέτρα. Και πιστεύω ότι η ειλικρίνεια που μας χαρακτήρισε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών είναι υψής της σημασίας. Για τα τιμολόγια. Σας είπα θα είναι ένα τέλος προοδευτικά μειούμενο και θα πληρώνει περισσότερο εκείνος που ρηπαίνει περισσότερο. Και οι εταιρείε που έχουν ένα πρότιμο Euro 5, Euro 6 ε, ως ε, δύναμη του κινητήρα έχουν απαλλαγή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στο μαθηματικό αυτό τύπο, στη φόρμουλα που φτιάξαμε, υπάρχει το κίνητρο αυτό της οικολογικής προσαρμογής. Και καλή είναι η λύση, αλλά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει και στο Συμβούλιο να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, κατάλληλη διαμόρφωση. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα earmarking, δηλαδή ε, δέσμευση ενό κονδυλίου για μια συγκεκριμένη χρήση. Θα καταλάβετε και θα δεχτείτε κι εσείς ότι για κάποιο ειδικό πρόγραμμα θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που μπορείς να το συγκεντρώσεις κατά 90-95%. Και απομένει τώρα γίνεται συζήτηση για το πώς θα μοιράσουμε τα χρήματα ή πού θα τα δαπανίσουμε. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι το σημαντικότερο εδώ είναι όχι τι χρώμα είναι η γάτα, αλλά πιάνει ποντίκια. Και ούτε μας νοιάζει το χρώμα του ποντικιού να είναι άσπρο ή μαύρο. Να το πιάσουμε θέλουμε και να πιάσουν τόπο και τα λεφτά μας. Ε, αυτό μας ενδιαφέρει και με κάποια συμμετοχή του εθνικού προϋβολογισμού. Ε, βεβαίως, κάποιες χώρες δυσκολεύονται πάρα πολύ και θα πρέπει να δούμε τι ε, γίνεται και ποια είναι τα προγράμματα, τα έργα, τα δίκτυα κτλ. και υποδομές. Και κάτι άλλο που θέλω να πω και το είπα και στο παρελθόν, έτσι και θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και οι προσπάθειές μας είναι να έχουν ύψη στην προτεραιότητα τα διευρωπαϊκά δίκτυα και μάλιστα ως προς τις μεταφορές TNT ε, και να συμφωνήσουμε Σε διάφορα κράτη-μέλη ε, λοιπόν ε, πρέπει να κάνουν προτάσεις και να πάρουν θέση και να τα γνωρίζουν αυτά και τα θεσμικά όργανα. Έγινε λοιπόν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, δεν έχει πρικοδοτηθεί 100% η νύφη, αλλά θα προσπαθήσουμε να λύσουμε και τα εναπομείναντα ζητήματα και με τον τρόπο αυτό να ε, προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Ένα άλλο στοιχείο που αναφέρατε είναι τα δικαιώματα των επιβατών. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να σας πω σχετικά με αυτό ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μην αναγνωρίζεται με αλφαγιώτα γενικά και όριστα η αρχή, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι στα δικαιώματα των επιβατών όταν υπήρχε κάποια πίεση από το Κοινοβούλιο και για τις οδικές μεταφορές και για τα λεωφορεία ε, για καλύτερη ρύθμιση η πρώτη ομάδα που αντέδρασε ήταν οι σιδηρόδρομοι οι οποίοι είπαν γιατί να δίνετε τόσα δικαιώματα στους επιβάτες των λεωφορείων, ενώ εμείς στο σιδηρόδρομο έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Και πριν να σας πω ότι ο πρώτος τριμερής διάλογος που έγινε μεταξύ της Προεδρίας, της Βελγικής προκειμένου ε, στο Κορεπέρ 1, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήταν πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού. Το λέω αυτό με κάποια χρονική απόσταση πλέον. Και χρειαστήκαμε πάρα πολύ ενέργεια και έμπνευση να δαπανίσουμε εκεί, ελπίζοντας να ε, επιτύχουμε ένα συμβασμό με κάποια ισορροπία σε αυτό το θέμα. Παράδειγμα. Στο Συμβούλιο χρειάστηκε ένα ορισμό στο τι εστί περιφερειακή συγκοινωνία, τοπική συγκοινωνία. Ε, εξαρτάται από την απόσταση και μόνο. Παράδειγμα, σε κάθε χώρα ο ε, ε, όρο και μόνο περιφερειακός ή τοπικός έχει άλλη ερμηνεία. Επίσης τα δύο συνοριακά. Θα επανέλθω στη συνέχεια σε αυτό. Γιατί υπάρχει η τοπικος εχει αλλη ερμηνεια επιση τα μικρή διασυνοριακή κυκλοφορία που έχει κάποια προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Γι' αυτό χρειάστηκαν κάποιες προσωρινές μεταβατικές ρυθμίσεις με εξαιρέσεις για να λυθούν προβλήματα και σε τοπικό επίπεδο και εντός των χωρών αλλά και σε χώρες που είχαν συμφωνίες διμερείς με χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις και το συνολικό πακέτο δικαιωμάτων των επιβατών και συγκεκριμένα των επιβατών με περιορισμένη κινητικότητα. Όλους ιδιαιτέρω που ενδιαφέρουν πάρα πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω τελικά θα μπορέσει να υπάρξει ένα συμβιβασμό, τουλάχιστον αυτό το ελπίζω. Αν ε, θέλετε για να σας <laughs> το ε, πω έτσι και προσπαθούμε να χαϊδεύουμε τώρα τους πάντες ε, να τους καλοπιάνουμε ε, για να δεχτούν τη συμφωνία χωρίς να μας χειροκροτεί κανείς ιδιαίτερος. Ε, βάζουν όλοι λίγο νερό στο κρασί τους για να περάσει γι' αυτό. Για στις μεταφορές γενικότερα προσπαθούμε να επιτύχουμε μια συμφωνία και στα δικαιώματα των επιβατών. Δεν θέλησαμε να επιβάλλουμε κάτι στις χώρες για να είναι όλοι δυσαριστημένοι και κανείς ικανοποιημένος. Τώρα, ε, για την οδηγία για τη διασυνορική κυκλοφορία σας είπα ότι έχουμε κάνει ήδη πολύ σημαντική πρόοδο. Ε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω εγώ εδώ ότι με τις διάφορες αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει κάθε χώρα ως προς τις παραβάσεις ε, που γίνονται στη οδική κυκλοφορία. Ε, είτε ασχολούνται με αυτά τα θέματα Υπουργεία Μεταφορών, η Δικαιοσύνη, το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέπει αστυνομία. Ε, βρήκαμε μια λύση όπου στο Κορεπέρ, στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων στις 15 Σεπτεμβρίου, ε, σχεδόν και επιτέλους θα έλεγα, συμφώνησαν επί της αρχής για τη νομική βάση το άρθρο 87 προκειμένου της συνθήκης. Και τώρα επιτέλους υπάρχει μια γνήσια προοπτική για μια καλή ρύθμιση. Και νομίζω ότι βάσει αυτής της συμφωνίας του Κορεπέρ μπορούμε να προχωρήσουμε ε, στις λεπτομέρειες και στη ρύθμιση των ζητημάτων. Κάποια ειδικά που με ρωτήσατε σε ό,τι αφορά την αυσιπλοεία και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στην Αυσιπλοεία, ΕΜΣΑ. Δεν ξέρω, μπορεί να σας φανεί ότι είναι δική μου παραξενιά αυτό, αλλά ε, ανέκαθεν υποστήριζα ότι ε, στις χερσαίες μεταφορές ε, στην Ευρώπη μας ενδιαφέρει πολύ η εσωτερική αγορά και έχουμε προωθήσει τις σχεσές μεταφορές, αλλά στην ακτοπλοεία δεν έχουμε καταφέρει με οικολογικό τρόπο να κάνουμε μεταφορές από τα θαλάσσια λιμάνια. Και την επιμελητία στα λιμάνια μας. Και αρμόδιοι για τα θέματα των οικονομικών και των τελωνίων δεν έχουν καταφέρει να συνοηθούν για μια διασυνοριακή ε, ακτοπλοεία για, για να μεταφέρονται έτσι τα εμπορεύματά μας. Στο άτυπο λοιπόν συμβούλιο ε, σας είπα ότι είχαμε ένα σύστημα blue belts και blue lanes έτσι λέγονται αυτά ε, στη γλώσσα την τεχνική και ε, από τη σκοπιά των τελωνίων και των οικονομικών ως προς τους ελέγχους συζητήθηκε γι' αυτό και καθημερινά ε, δεν θέλαμε να αποφεύγουμε τις καθημερινές επικαλύψεις, επαναλήψεις και με την έμσα για να έχει ένα έλεγχο και μια παρακολούθηση και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη στιγμή έχει γύρει ένας τελωνιακός έλεγχος σε κάποια από τις χώρες ε, να είναι δεδομένη ασφάλεια ότι δεν χρειάζονται άλλοι έλεγχοι ε, για να σταματήσουν τα διοικητικά εμπόδια και όχι σε κάθε λιμάνι να ελέγχεται από το τελωνίο. Κάναμε μια δοκιμή, ε, ε, εγκρίναμε τη δοκιμή αυτή και τελικά ελπίζουμε ότι θα είναι θετικό το αποτέλεσμα. Έτσι ώστε και η εκτοπλοεία θα μπορέσει να συμπεριληφθεί και στις εμπορευματικέ μεταφορές για να αποσυμφορηθούν και οι αυτοκινητόδρομοι στην Ευρώπη. Με μεγαλύτερη συμμετοχή της παράκτειας, επαναλαμβάνω, ναυσιπλοίας, της ακτοπλοείας. Τώρα για τη ρήπανση και ε, αυτά που αναφέρατε για τις εκπομπές θείου ας πούμε και ε, τα θέματα της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας από τη μια και τη Μεσογείου από την άλλη πρέπει να σας πω ότι ο συμβασμός που πετύχαμε εκεί είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε και βασίζεται στην πολιτική ε, πραγματικότητα. Σε ορισμένα μέρη της Υπήρου μας υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προθυμία από ό,τι σε κάποια άλλη. Ε, προσπαθούμε και οικολογικά, ε, από πλευράς ε, περιβάλλοντος δηλαδή, να πετύχουμε το εφικτό. και να κάνουμε πιο αυστηρούς κανόνες για τις ρυθμίσεις για να προχωρούμε και προς την περιβαλλοντική αυτή κατεύθυνση. Να σας πω και ένα μικρό περιστατικό, έτσι, ανέκδοτο για την υπέρπτυση της Σιβηρίας. Ο Σλοβάκος συνάδελφος νομίζω το ρώτησε αυτό. Ε, θα ήθελα να πω ε, ότι έχουμε διμερείς συνομιλίες Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσική Ομοσπονδία Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κύριος Κάλλας ήδη απίφθινε μία έκκληση για εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας και όχι να αναβληθεί όπως ζητούν κάποιοι άλλοι. Αλλιώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προσφυγή επί παραλήψη ή παραβίαση της συνθήκης. Πάντως πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να ε, συζητήσει με τη Ρωσία αυτά τα θέματα. Πρόεδρε, νομίζω ότι τελείωσα, απάντησα, δεν ξέρω αν χρειαστεί να προχωρήσουμε. Uh, Ωραία. Ε, να ακούσουμε τώρα τις ε, ερωτήσεις. Η πρώτη κυρία Ριβέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βελγική Προεδρία για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση των δραστηριοτήτων του πρώτου τριμήνου Χαίρομαι που μπόρεσε να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών για την οδηγία Ευρωμηνέτα που επέτρεψε σε αυτό σημαντικό για να προχωρήσει. Σήμερα οργανώνεται μια Ευρωπαϊκή Συνάντηση Κορυφής τη Αεροπλοεία στην ε, Μπρίζ και υπάρχει απουσία ευρωβουλευτών. Αντίθετα βλέπω ότι στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται μια συνάντηση για τους ενιαίους για τους ουρανούς, η συνάντηση αυτή έθεσε ως προτεραιότητα την δημιουργία των ε, ενιαίων ουρανών. Η έκρηξη του Ισλαδικού Ισβεστίου έδειξε ότι πραγματικά αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχει σκοπό να συμβάλει η Βελική Προεδρία σε αυτό το στόχο επιταχύνοντας την εφαρμογή των ενιαίων ουρανών. Ευχαριστώ, κύριε Λάιτρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Εμένα με απασχολεί μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει και το Συμβούλιο στο μέλλον. Ε, πρόκειται για μια έκθεση που εκρεμεί εδώ σε που ε, ε, έκθεση Πασκάλη για την ασφάλεια των αερομεταφορών, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων το να εισαχθούν σαρωτές σώματος στα αεροδρόμια. Αυτό που με απασχολεί είναι το εξής. Πριν λίγο καιρό, υιοθετήθηκε στο Κοινοβούλιο μια έκθεση που είχε να κάνει με την ε, χρηματοδότηση των μέτρων ασφαλείας στα αεροδρόμια. Και δεν αναφέρατε στην εισαγωγή σας ε, την ε, πρόταση αυτή. Προφανώς επειδή το Συμβούλιο δεν έχει πολλά να πει για αυτήν. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν γίνεται τίποτα στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Θα θεωρούσε κανείς ότι το πρόβλημα είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτό, αλλά εάν υποθέσουμε ότι συζητιέται η, μία η έκθεση για ε, την ασφάλεια χωρίς να συζητιέται το πώς θα χρηματοδοτηθεί. Μπορεί να αποτύχει η πρόταση αυτή. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν Ποια στρατηγική έχετε, τι στρατηγική έχετε για να προωθήσετε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο, ώστε να έχουμε καλό αποτέλεσμα και από τις δύο αυτές εκθέσεις. Ευχαριστώ κύριε Λάιχτφριντ, η κυρία Λίχτεμπεργκερ, δύο λεφτά. Ευχαριστώ θερμά. Καταρχήν να επενέσω την Βελγική Προεδρία, διότι ε, έχει αναλάβει ε, πρωτοβουλίες σε θέμα το οποίο πολλοί απέφευγαν επειδή το θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο. Δυστυχώς το αποτέλεσμα για χώρες στο κέντρο της Ευρώπης που ε, ε, φέρουν ε, μεγάλο μέρος των μεταφορών. Ε, ο συμβιβασμός αυτός δεν είναι ικανοποιητικός. Λέμε ότι πρέπει να πιάσουμε το ποντίκι και κατόπιν να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Αλλά στα δικά μου μάτια πρόκειται για ψήλο. εάν υπολογίσουμε αυτά που έχουν αποφασιστεί, τότε όλα, ε, αν τα υπολογίσουμε με βάση τα 100 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Και εάν θέλουμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα, έχω αμφιβολίες. Διότι τουλάχιστον ξέρω την αριθμητική των τεσσάρων πρώτων τάξεων του σχολείου. Πιστεύω ότι αν δεν είμαστε πιο φιλόδοξοι, ή τουλάχιστον εισάγουμε σχετική υποχρέωση, τότε η ευρωβινιέτα δυστυχώς θα παραμείνει συμβολική. Δεν θα είναι τελείως άνευ σημασίας, διότι τουλάχιστον αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν ε, οι οικολογικές δαπάνες, αλλά δεν θα ε, σημάνει μεγάλη διαφορά. Ε, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Εάν δεν θέλουμε να γίνουμε ρεζίλοι στους πολίτες της Ευρώπης, τότε δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο να επιτρέψουμε ε, ένα σωρό παρεκκλήσεις. Σας παρακαλώ αυτό να το λάβετε υπόψη σας. Επίσης, όσον αφορά τη σύμβαση των Άλπαιων, παρακαλώ να απαντήσετε. Ήδη τέθηκε η ερώτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεγκράντης Πασκουάλ. Μάλιστα. Θα ήθελα καταρχάς να επενέσω και να εκθιάσω τη Βελγική Προεδρία που αποδεικνύει ότι άλλη, άλλη μια φορά ότι η φαινομενική αστάθεια και ο εύθραυστος χαρακτήρας μπορεί να συνοδεύεται από μια πολύ στιβαρή προεδρία. Ο κύριος Σίμψον δεν μου δίνει ε, ε, άλλο χρόνο για επένους. Όπως γνωρίζετε, θα περάσω τώρα στην κριτική, όπως γνωρίζετε η Ισπανία είναι κατά της Ευρωβινιέτας. Είναι ε, αποτυχία. Δεν ε, ε, εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των μέσων ε, μεταφοράς. Δεν είχε το θάρρος η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει τα λιμάνια και να έχουμε αυτές τις λεωφόρους, τις θαλάσσιες. Και η χώρα μου, όπως και άλλες, ε, σύρθηκε στα δικαστήρια γιατί δεν εφαρμόζουμε σωστά το πακέτο των σιδηροδρόμων και στο μόνο που τολμάμε κάτι να κάνουμε είναι ο καημένος αυτοκινητόδρομος για να λειτουργεί και αγορά. Στις 6 Οκτωβρίου πετύχατε μια συμφωνία που είναι πιο θετική από τα προηγούμενα, εντάξει, βελτιώνει πια ποια πράγματα και αυτά που ορισμένοι μπορούν να τα θεωρούν αρνητικά. Εγώ τα θεωρώ θετικά. Μας δώσει χρόνο κύριο Σίμψον, μπορώ να αναφέρω και τα θετικά. Πάντως η Ισπανία δεν μπόρεσε να το δεχτεί γιατί ε, είναι επιβαρυντικό για μας και διακριτική μεταχείριση και για άλλες περιφερειακέ χώρε που στην Ευρωβινιέτα δεν βλέπουμε κανένα όφελο. Και λέει θα είναι στους αυτοκινητοδρόμους αυτό και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Εντάξει. Καλό αυτό. Θα πρέπει το Συμβούλιο να υποστηρίξει έστω και ε, με μέρη την πρόταση του Κοινοβουλίου να εξαιρούνται τα ε, οχήματα που είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικά. Και επίσης οι ώρες εχμής ρυθμίστηκαν με τρόπο καλύτερο από αυτό που ελπίζαμε. Πάντως, ε, χαιρόμαστε για τη διαφάνεια αυτή της απόφασης τη 6 ε, Οκτωβρίου, αλλά η Ευρωβινιέτα για μας δεν φαίνει τίποτα θετικό στη διαλειτουργικότητα και στις συνδυασμένε μεταφορές και θα μείνει όρνος, όνειρο θε, θερινής νυχτός για να μην πω χρονικό προαναγγελθέντους θανάτου. Η Τσεχία ε, ακολούθησε άλλη προεδρία, μετά ε, η Ισπανία, τώρα ε, το Βέλγιο. Πραγματικά είναι αυτό το θέμα και το πασάρι η μια προεδρία στην επόμενη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Α, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Γίνεται μεγάλη αναφορά τον προγραμματισμό, περιορισμένη αναφορά στην εφαρμογή, στην πραγματοποίηση, στο timing. Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μερικών υποδομών. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Ήμουν σε μία διπλανή αίθουσα και δείξαμε το θέμα της καινοτομίας. Η καινοτομία και οι υποδομές είναι οι δύο βασικοί τομείς που ενδεχομένως θα μας βοηθούσαν να ξεπεράσουμε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο ή τρία θέματα που έθιξαν μερικοί συνάδελφοι, το δικαίωμα των επιβατών. Ήρθατε σε τρει τριμερεί διαλόγου. Στον πρώτο δεν είπατε τίποτα, στο δεύτερο είπατε 500 χιλιόμετρα, εφαρμοστέω σε πέντε χρόνια. Δεν ξέρω, με συγχωρείτε κατά την άποψή σα, αυτό σημαίνει ε, κατά πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια σε ό,τι αφορά την ευρωμηνέτα Εγώ έχω ορισμένε αμφιβολίε. Αυξάνουμε τι ε, τιμέ ε, για άλλα μέσα μεταφορά, αλλά δεν δημιουργούμε τι απαραίτητε προποθέσει προποθέσει για να αναπτυχθούν άλλα μέσα μεταφορές. Θέλουμε να πληρώσει ο χρήστη την. Ε, ε, τη, τη ρήπανση, ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν να πάρουν το Eurofed. Θέλουμε να ε, πληρώσει την ε, συμφόρηση αυτός που την υφίσταται. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ. Δεν μιλάμε πια για δημόσιες μεταφορές. Μιλάμε για ένα equity που συν, που στην ουσία διακυβεύει τα όσα αποφασίστηκαν προηγουμένως. Προσοχή λοιπόν να στα δούμε αυτά τα προβλήματα γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο επικίνδυνο όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα. Δύο ε, ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Δύο ερωτήσεις έχω για την Ευρωβινιέτα. Μιλήσατε για τις ε, δαπάνες συμφόρησης και είπατε ότι έχει βρεθεί ισορροπημένη λύση. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ισορροπημένη λύση αυτή. Μήπως μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό σύντομα. Και δεύτερον, πιστεύετε προσωπικά πράγματι ότι ε, χωρίς ε, να, ε, εάν δεν ε, προορίζονται οι, τα χρήματα της Ευρωβινιέτας για συγκεκριμένους σκοπούς θα μπορέσουμε να πετύχουμε μείωση των, των εκπομπών. Αν συμφωνείτε θα παραβιάσω τις αρχές μου και θα σας επιτρέψω να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε να μας επισκεφτείτε δεν είχα σκοπό να θέσω την ερώτηση αυτή. Ήλπιζα ότι το θέμα αυτό που ήδη ετέθη θα είχε απαντηθεί με έναν τρόπο πιο συγκεκριμένο. Η ερώτησή μου αφορά τα καύσιμα της ναυσιβλοίας. Τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση. Ξέρω ότι η Εστονία και η Φιλανδία δεν έχουν ε, ενταχθεί στο ΜΑΡΠ λέξη. Δεύτερη ερώτηση. Δεν αναφέρατε ότι οι δύο αυτές χώρες που ήταν οι τελευταίες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παροχημένα μεταφορικά, συστήματα μεταφορών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διευρωπαϊκά συστήματα μεταφορών αν δεν ξέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τελειώσαμε. Θα δοθούν ε, απαντήσεις. Ελπίζω μέσα σε 9 λεπτά να τα καταφέρετε κύριε Υπουργέ. Το πρώτο για το SIS, Single European Sky. SIS. Ε, αγνοώ κυρία μου τι έγινε χτες, πραγματικά αγνοώ για τον ενιαίο ουρανό. Δεν συμμετείχα εγώ σε εκείνη τη συζήτηση, αλλά από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει χαλάσει με το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω. Ή το Κοινοβούλιο με την Επιτροπή. Δεν επικοινωνείται πλέον. Γιατί ως συμπέρασμα μου είπε ο κύριος Κάλα σήμερα το πρωί ότι ε, σκέφτεται να κάνει νέα πρόταση στο Συμβούλιο για να προσπαθήσει να ε, βγει ε, από τη θέση αυτή. Αποσύρει την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί λέει δεν την έκανα δεκτή, την αποσύρω, κάτι άλλο πρέπει να κάνω για να κουνηθούν. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δυστυχώ από αυτού δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πρέπει να περιμένω. Δεν θα προσπαθήσω γιατί σήμερα το πρωί μόλι πήρα αυτή την πληροφορία, θα πρέπει να ενημερωθώ και ο ίδιο να δω τι συνέβη και να προσπαθήσω να, να καταλάβω τον προσανατολισμό που θέλει μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Βέβαια, σε αυτό το θέμα του νέου Ευρωπαϊκού Ουρανού 2, ε, κάνουμε εμείς κάποιες προσπάθειες και οι Βέλγοι και στα πλαίσια του ΦΑΜΠΕΚ. Θα κάνουν μια συμφωνία στο εσωτερικό λοιπόν για τον Μπενελούκ στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία και θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι το μεγάλο θέμα στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εμεί θέλουμε να κάνουμε πρόοδους, διότι θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον των εναέριων μεταφορών να υπάρξει συμφωνία μεταξύ της πολιτικής και της ε, πολεμικής αεροπορίας για να υπάρχει και μια καλύτερη διαχείριση και πολύ πιο οικονομική του συνόλου των δραστηριοτήτων της ενέργειας κυκλοφορίας. Επί της αρχής λοιπόν, ελπίζω οι πάντες να παραμείνουν πεπισμένοι ότι χρειάζεται κοινή διαχείριση και ε, πολιτικές λοιπόν, και ε, ε, στρατιωτικές μεταφορές σε αέριες μεταφορές Κυρίως η πολιτική αεροπορία να μην ε, υφίσταται τις συνέπειες της πολεμικής αεροπορίας. Αλλά αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, είμαι ανίκανος να σας δώσω τον προσανατολισμό. Θα πρέπει να συζητήσω, να συνοηθώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δω προς ποια κατεύθυνση θα βαίνει μια ενδεχόμενη νέα πρότασή της. Χίλια συγγνώμη και πάλι, αλλά τι να κάνω δεν θα μπορούσα να σας ενημερώσω περισσότερο. Για τους αρωτές σώματος στα αεροδρόμια και την έγκριση. Στην Μπρουζ συζητούμε με όλους τους ενδιαφερομένους για την εναέρια κυκλοφορία και τους ενεχομένους και αυτό το θέμα είναι επιτάπητος. Ο άλλος κύριος έφυγε. Α, όχι, εδώ είναι. Για αυτό το θέμα γεγονός είναι ότι για τους ερωτές σώματος, ανεξάρτητα από τη φόρμουλα και τη λύση που θέλουμε να εφεύρουμε και να εφαρμόσουμε, είναι γεγονός ότι επιμένουμε σε μια λύση που να είναι αποτελεσματική από πλευράς τεχνικής και τεχνολογικής, να επιτρέπει να αποφεύγουμε τις φορές που βλέπουμε σήμερα και από πλευράς επίσης δημόσιας υγείας να σέβεται απολύτως τη δημόσια υγεία και να μην είναι περισσότερα τα μειονεκτήματα από τα πλεονεκτήματα σε αέριες μεταφορές. Και να μην είναι σε μειονεκτική θέση αέριες μεταφορές σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς που δεν χρειάζεται τέτοιου ελέγχους. Και πάλι ε, είναι δηλωμένη ε, η βούλησή μας και η πρόθεσή μας. Αλλά η καλή πρόθεση και η καλή βούληση δεν είναι κάτι που κατά κανόνα βλέπουμε ε, στις ομάδες των διαφόρων ε, φορέων που διαχειρίζονται τα αεροδρόμια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύμβαση των Άλπαιων. Ε, κάθε φορά το βρίσκω μπροστά μου αυτό. Ε, ξέρετε τι, ωραία είναι να αναφέρουμε κάπου τέτοια θέματα και να τα παραπέμπουμε στην Προεδρία, αλλά στη σύμβαση των Άλπαιων θα πρέπει οι ενεχόμενοι φορείς, τα συμβαλόμενα μέρη να έχουν την πρόθεση να προχωρήσουν σε μια συμφωνία. Τι να σας κάνω. Γνωρίζω ε, τι λέει η μία χώρα, οι μερικές χώρες που στρέφονται κατά άλλων, αλλά αν έχουμε ως αφετηρία ότι ε, ε, υπάρχει πλήρη απροθυμία από πλευράς ενός βασικού εταίρου, Εμεί τι να κάνουμε ως Βελγική Προεδρία για να το λύσουμε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε ε, μόνοι μας να κινήσουμε την κατάσταση αυτή, αν δεν υπάρχει βούληση. Ειδικά για τη σύμβαση των Αλπαίων υπάρχουν ειδικά προβλήματα που αφορούν τις συγκεκριμένες χώρες και ρώτησε κάποιος που μάλλον από την Αυστρία κατάγεται από ό,τι κατάλαβα. Τι γίνεται με τα ειδικά προβλήματα. Να σας πω για την Ευρωβινιέτα. Να σας διαβάσω και το κείμενο αν θέλετε που εγκρίθηκε. Ε, οι τιμές του πίνακα 1. Ο πίνακας 1 είναι η τιμολόγηση ε, ανάλογα με τους διάφορους κινητήρες Euro 0 κτλ. φτάνει μέχρι δύο σε ορεινές περιοχές στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται από την κλίση ε, το, ε, του, του, δρόμου, ε, τη θερμοκρασία και κάποιους άλλους παράγοντες. Αυτά πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που ζητήθηκε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς την κατάσταση. Ε, ο πολλαπλασιαστή, ο παράγων είναι 2, δεν είναι 3 ή 4, αλλά είναι πάντω αύξηση. Δεν μπορούμε να ζητάμε και το ανέφεκτο γιατί δεν θα πετύχουμε τίποτα. Θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Για την Ευρωβινιέτα και τις διαφορές και τις διαφωνίε, θα είπε ο κύριο Γκράντε. Κοιτάξτε, το είπα νομίζω και στην εισαγωγή μου. οι περιφερειακές χώρες της Ευρώπης έχουν τελείως διαφορετική θέση από τις κεντρικές χώρες της Ευρώπης. Και γεωγραφική αλλά και τοποθέτηση. Για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία χρειάστηκε να βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους. Το είπα και πριν. Παράδειγμα. Υπήρξαν κάποιες περιφέρειες, ε, ζώνες που έχουμε την υψηλή ταρίφα, που είναι 175% του βασικού, ποσού και εκεί λήφθησαν υπόψη διάφορες ε, ε, απόψεις χωρών όπως και η δική σας. Αλλά είπαμε σε ώρες ε, που είναι άδεια αυτοκινητόδρομη να είναι χαμηλότερα τα τέλη αυτά και χαμηλότερο το βασικό ακόμα. Συμβασμός κύριε Ντεγκράντες ξέρετε ότι εξορισμού μένουν όλοι δυσαρεστημένοι. Αλλά και όλοι έχουν καταφέρει να περάσουν ορισμένα από τα αιτήματα ή τις απαιτήσει τους. Αυτό είναι ο συμβιβασμό. Δηλαδή έχει και λίγο κρασάκι μέσα. Παρόλο που ε, είναι πολύ το νερό. Ε, έχει και λίγο κοκκινούλι, λίγο κίτρινο αν είναι λευκό το κρασί και έχει και γεύση κρασιού ελαφρώς όσο νερό και αν βάλαμε. Τι άλλο με ρωτήσατε. Ε, για την περιεκτικότητα σε θείο. Όταν παίρνει αποφάσεις ο ΑΕΜΟ, ο Διεθνής ε, Οργανισμός που ενδεχομένως, ενδεχομένως λέω και το λέω προσεκτικά, ε, δεν τα έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά και βάζει πολύ αυστηρούς κανόνες, δηλαδή από την πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο την κάνει σχεδόν μηδενική, τότε ε, κινδυνεύουμε να καούμε. Τελικά, τι βγήκε, το 0,1 ως τιμή είναι πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ αυστηρό και επηρεάζει οπωσδήποτε την οικονομική ζωή όλων των ε, ε, εταιριών αυσιπλοίες που έχουν ε, να λύσουν αυτό το ζήτημα πολύ πιο ρεαλιστικό θα ήταν σε μια πρώτη φάση να πάμε στο 0,5. Αλλά μην ζητάτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, να λογοδοτήσει για αποφάσεις που έχει πάρει ο Διεθνής Οργανισμός για την Αυσιπλοεία. Έχοντας πλήρη γνώση των πραγμάτων και το έχει πάει εκεί. Θα προσπαθήσουμε, και αυτό θα είναι και ε, καθήκον ε, διαφόρων κρατών, θα προσπαθήσουμε, λέω, να ε, πιέσουμε και να καταλάβουν ότι θα πρέπει να μπει κάποιο χρονικό ε, περιθώριο για να αφαιρεθεί ακόμα περισσότερο το θείο από τα καύσιμα των πλοίων και να μην αρχίσουν να πέφτουν τώρα τα αυστηρά ε, αυτά πρόσημα. Γιατί θέλουμε κανόνους, κανόνες παιχνιδιού ίδιους για όλους και στη θάλασσα Και αυτό είναι αρνητικό για ε, εταιρείε της βορειοδυτικής Ευρώπης, ας πούμε, σε σχέση με άλλες χώρες που δεν θα το τηρήσουν αυτό παρά τους κανόνες του IMO σε διάφορα ύδατα που δεν θα μπορούν να ε, ταξιδεύουν και ύδατα ε, χωρικά δικά μας. Τα γνωρίζουμε αυτά. Και για τη Βόρεια Θάλασσα και για τη Βαλτική ισχύουν άλλα πρότυπα και άλλα στάνταρτς και οι χώρες που βρέχονται από τις άλλες αυτές έχουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις, αλλά αυτό το βήμα που έκανε ο ΑΕΜΟ νομίζω ε, ήταν υπερβολικό ε, και επιβαρύνει πάρα πολύ την οικονομία και τη ζωή των επιχειρήσεων. Το πρότυπο τώρα για το θείο λοιπόν την περιεκτικότητα του καυσίμου των πλοίων θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα στι περισσότερε ερωτήσει έτσι δεν είναι. Α, ναι, ναι, κάτι που ξέχασα. Για τι υποδομέ και την κατασκευή νέων υποδομών. Ποιο ρώτησε, ο κύριο Καντσιάν. Τα νέα έργα υποδομών. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν είναι στα χέρια μου, τα δικά μα. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει λίστα προτεραιοτήτων για τις συνδέσεις που λείπουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. Και κάθε χώρα θα πρέπει να επιδείξει αρκετό ευρωπαϊκό πνεύμα για να τα δεχτεί αυτά. Αλλά ας κάνει αυτή την απογραφή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά με τη δέσμευση αυτών των κονδυλίων, με το earmarking, να δούμε αν υπάρχουν τα κατάλληλα κονδύλια και όταν τα βρούμε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα κατά προτεραιότητα υπερεθνικά. Ο χρόνος μας πιέζει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα μας είπατε. Θα ήθελα όμως ε, να σας ευχαριστήσω ως Προεδρία που εμπλέξατε το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Μεταφορών σε πολλές από τις πρωτοβουλίες που λάβατε κατά τη διάρκεια των άτυπων συναντήσεων του Συμβουλίου. Πραγματικά εκτιμάμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες που καταβάλατε να μας συμπεριλάβετε στους προβληματισμούς σας. Προσωπικές ευχαριστίες λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας επιτρέπουμε τώρα να επιστρέψετε στην Βρύζ και να μιλήσετε για την αεροπλοεία. Ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι συντονιστές σε λίγο.